ποτέ να τα

Καλημέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ την κυρία Σπινόσα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ισπανίας. Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2010. Αυτή τη στιγμή τίθεται σε εφαρμογή η συνθήκη τη Λισαβόνα, που σημαίνει ότι θα αλλάξει ο τρόπο λήψη αποφάσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και θα έχουμε και μεταρρύθμιση κοινή ελευτική πολιτική και μα χαροποιεί λοιπόν το γεγονό ότι αλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα με μακρά αλλιευτική παράδοση που θεωρούμε ότι θα δώσει ε, τη δέουσα προτεραιότητα στα θέματα που θα μας αποσχολούν. Τα θέματα τα οποία θα αποτελέσουν προτεραιότητα είναι πολύ εύκολο να τα εντοπίσουμε. Σε νομοθετικό πλαίσιο θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθετική διαδικασία, την ε, διαδικασία σε προτάσεις οι οποίες είναι σε εξελίξη αυτή τη στιγμή, κυρίως και την εφαρμογή του κανονισμού Omnibus, τον οποίο διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και το θέμα της εποπτείας, το οποίο ε, είναι θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χθε στη συνεδρίαση των συντονιστών λάβαμε και τι δέουσε αποφάσει. Σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Θα έχουμε τα αποτελέσματα τη διαβούλευση η οποία μόλι ολοκληρώθηκε μεταξύ κρατών μελών ε, ε, Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των ενδιαφερομένων για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση για τις προσανατολισμούς στους οποίους θα πρέπει να βασιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση των μελλοντικών προτάσεών όσον αφορά τώρα τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων είναι λίγο ιδιαίτερη η περίοδος αυτή διότι θα χρειαστούμε μια περαιτέρω προσπάθεια προσαρμογής. Το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί μια πραγματική ε, και όσο το δυνατόν ε, στενότερη συνεργασία σεβόμενη το γράμμα της συνθήκης. Σε όλους τους τομείς της αλίας και της γεωργίας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προασπίσουμε το αλλιευτικό περιβάλλον και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς επίσης και τους πολίτες μας. Αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει ε, τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, όπως και στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες αποκαλούμε τρίλογο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να ελέγχει τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία διαπραγματεύεται τις διεθνείς συμβάσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα να πω ότι επειδή υπάρχει ισοτιμία ρόλων πλέον μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, κατά την προετοιμασία για τις κοινέ θέσεις, ε, για τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας και ε, να δούμε και τι γίνεται με τις αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Έχουμε ήδη γνωστοποιήσει τη θέση μας στην υποψήφια επίτροπο την κυρία Δαμενάκη στην ακρόαση η οποία έγινε στο Στρασβούργο και τις επαναλαμβάνουμε και σε εσά, κυρία Υπουργέ με στόχο στο μέλλον να, υπάρχει, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία επί του θέματος. Μετά από την αρχική σας παρέμβαση την οποία υπολογίζω ότι θα κάνετε σε 20 λεπτά περίπου, αλλά φυσικά εσείς έχετε την ευελιξία που δίνουμε πάντα στις ε, προεδρίες. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και στη συνέχεια μπορούν να παρέμβουν όλοι οι ευρωβουλευτές, σεβόμενοι πάντα και το χρονοδιάγραμμα της ε, Υπουργού. Κύριε Υπουργό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω ότι η Προεδρία ε, δεσμεύεται, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Σαπατόριο στην ε, ε, παρέμβασή του στην Ολομέλεια, να συνεργαστούν στη διάρκεια όλου του εξαμήνου σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλους εσάς. το είπε και η πρόεδρος στην παρέμβασή της, αναφερόμενη στις αλλαγές οι οποίες έχουν προκύψει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ε, πράγματι, ε, μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, αυτή η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι τα θέματα που μας απασχολούν θα προχωρήσουν δεόντως και ε, εάν υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Πριν περάσω στις λεπτομέρειες για το πρόγραμμά μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια ε, για να ευχαριστήσω τα όσα έκανε ο προκάτοχός μου, ο Υπουργός Εσκίλ Ερλάνσον. Τόσο η οθέτηση του νέου κανονικού, κανονισμού εποπτείας, όπως επίσης και η έγκριση του νέου κανονισμού τάκ και ποσοστώσεων για το 2010, ήταν αποτέλεσμα του επαχθούς ορισμένες φορές έργου που χρειάστηκε να ε, ολοκληρώσει η Σουηδική Προεδρία. Μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτής της Προεδρίας, τις οποίες θα σας παρουσιάσω τώρα και θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομη για να ε, μπορέσουμε να έχουμε και χρόνο να συζητήσουμε για να μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που θα θέλετε να μου θέσετε. Όπως σας έλεγα λοιπόν, θα σας διαβιβάσω τώρα τις προτεραιότητες της Προεδρίας, οι οποίες θέλουν να προχωρήσουμε στον καθορισμό των αξώνων στους οποίους ε, θα βασιστεί η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Θα ασχοληθούμε επίσης με τρία πολύ σχετικά θέματα. Τη μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς, τα πολιετή σχέδια για το γάβρο, το σαβρίδι και το ε, βακαλάο του Ατλαντικού και επίσης την οικολογική επισήμανση των αλληλευτικών προϊόντων. Όσον αφορά τώρα στη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής, η διαδικασία προχωρά με καλούς ρυθμούς. Εχθές ε, ολοκληρώσετε και εσείς τη συζήτησή σας και την ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή σας. Ξέρω ότι είχαμε περίπου 400 ε, τροπολογίες, μπορεί και παραπάνω και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό θεωρείτε εσείς πόσο σημαντική θεωρείτε εσείς την Πράσινη Βίβλο και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και την ε, κυρία Πατάο Νέβες για την έξοχη δουλειά της. Μετά από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα περάσουμε στη συζήτηση στα πλαίσια του Συμβουλίου με στόχο να έχουμε ένα πολιτικό κείμενο φέτος. Κάποιοι θεωρούν ότι το να εφαρμόσουμε με επιτυχία την κοινή αλληλευτική πολιτική είναι μία αδύνατη αποστολή. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και θα θέλαμε να αναλύσουμε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει το θέμα της διατήρησης των ε, ε, αλλιευτικών αποθεμάτων και καθώς επίσης και το θέμα της ε, συμπερίληψης του περιβάλλοντος και της ναυτιλίας στην μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς, η αναθεώρηση της διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, καθορίσει τις απόψεις της, της μεταρρυθμίσεως αυτής και για την Προεδρία μας η συζήτηση θεωρείται ε, και απαραίτητη αλλά και κατεπίγουσα και θα πρέπει να γίνει από συνολική άποψη για όλα τα ληφτικά και προϊόντα και τα προϊόντα ηχθειοκαλλιέργειας και με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Όσον αφορά τώρα τα πολιετή σχέδια για συγκεκριμένα αποθέματα, ε, που είναι η τρίτη μας προτεραιότητα, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της μορφής ε, της διακλάδωσης ε, και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ορίζοντας διαχείρισης μακροπρόθεσμα, ο οποίος επιτρέπει στον κλάδο να προγραμματίσει τις δραστηριότητές του και να μην έχει αμφισημίες. Προγράμματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Εάν η Ευρώπη ήταν αυτή η οποία ήταν είχε τα ενία της καταπολέμησης παράνομης άναρχης και λαθρέας αλληλείας, ε, δεν θα πρέπει τώρα να σταματήσει στη διαχείριση των ελευτικών αποθεμάτων. Το θέμα του Γαύρου ε, είναι πρώτο στον κατάλογό μας. Να σας υπενθυμίσω στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αποφασίστηκε μετά από πολλά χρόνια να ξανανοίξει ε, η αλληλεία αυτού του είδους. Ισχύει ο κανονισμός ελέγχου ήδη και επομένω η συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εστιάσει στου ε, κύριους προσανατολισμούς και στη μελέτη για να καθορίσουμε το μέγιστο επιτροπήμενο αλίευμα όταν δεν έχουμε κατάλληλες πληροφορίες ε, και θα χρησιμοποιήσουμε την αρχή της πρόληψης. Όσον αφορά το Σαβρίδι, νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη μας ε, κοινή επιτυχία. Θα πρέπει να καθορίσουμε τις ζώνες διαχείρισης, αυτός είναι ο πρώτος στόχος που έχουμε και ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέσω ενός ή δύο άτυπων ε, τριμερών συναντήσεων. Τώρα, για το βακαλάο του Ατλαντικού έχει σταθεροποιηθεί ε, το απόθεμα και μπορέσαμε να καθορίσουμε ε, μια αύξηση για το ΤΑΚ ε, το συγκεκριμένο το Δεκέμβριο, γεγονό που χαροποίησε τους αλληλείς και θεωρούμε ότι ε, ο βακαλάος του Ατλαντικού θα πρέπει να παραμείνει ένα βιώσιμο απόθεμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει η πρόταση θα εξαρτηθεί και από την επιστημονική αξιολόγηση η οποία θα γίνει το Μάιο συγγνώμη το Μάρτιο και ε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πρόημο να σας πω οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο από τα θέματα τα οποία σας ανακοίνωσα είναι η οικολογική επισήμανση των αλευτικών προϊόντων. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος καταναλωτής παγκοσμίω αλευτικών προϊόντων. Είπαμε πώς μπορούμε να έχουμε βιώσιμη αλίευση. Επίσης θα ήθελα κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας να σκεφτούμε και τους καταναλωτές. Η θέση σε ισχύ του κανονισμού θα ε, επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν όταν το επιθυμούν αλλιεύματα τα οποία έχουν αλλιευθεί με βιώσιμο τρόπο και οι αλλιείς θα μπορούν από πλευρά τους να αποδείξουν ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλιεύουν υπεύθυνα. Εγκρίνοντα τον οριζόντιο κανονισμό, στόχος μας είναι να εστιάσουμε τη συζήτηση ε, στα όσα αφορούν την αλληλεία συγκεκριμένα. Θα αναθεωρήσουμε την κατάσταση της πρότασης στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο το Μάιο. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε δύο ακόμα θέματα. Το πρώτο είναι το σύστημα τεκμηρίωσης των αλλιευμάτων για τον τόνο Ξέρω ότι έχετε ετοιμάσει την, ετοιμάζετε την ε, ψηφοφορία ανατολισμού και θα είναι απαραίτητο για μας ε, και για σας να λάβετε υπόψη και ό,τι συμφωνήθηκε στο Ρεσίφε το Νοέμβριο του 2009 στην ε, ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού. Αυτό θα μας επιτρέψει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Διεθνών Οργανώσεων. Το δεύτερο είναι η τροποποίηση των απαιτήσεων πρόσβασης για τα ε, ψάρια βαθέων υδάτων. Ο κανονισμός χρονολογείται από το 2002, γι' αυτό και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα θέματα της πρόσβασης των πληροφοριών για την αλληλευτική προσπάθεια, καθώς επίσης και τα θέματα ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Να αναφερθώ τώρα στις εξωτερικές σχέσεις ε, στα πλαίσια της αλληλείας. θα πρέπει να σκεφτούμε και το διεθνή χαρακτήρα που έχει η αλία και κυρίως ε, για συγκεκριμένα λευτικά αποθέματα όπως είναι για παράδειγμα τα αλλιευτικά αποθέματα τα οποία είναι ε, πόροι που αγνοούν τα ε, σύνορα και ε, εξαρτούνται, εξαρτώνται από κοινά αλλιευτικά υποσυστήματα. Οι συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για τη διατήρηση της δραστηριότητας του στόλου μας και για να μπορέσει να είναι επαρκή η κοινοτική αγορά η οποία είναι η πρώτη στον κόσμο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την άμεση και έμεση απασχόληση σε θέματα λίας ε, και του κλάδου. Ε, η υπογραφή με τη Χιλή μια συμφωνίας για το Ξηφία ε, στην, νοτιοανατολική, στο νοτιοανατολικό ειρηνικό θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση του είδου. Στην περίπτωση της Μικρονησίας και του Σάντο Τομέι Πρίνσιπε, το Συμβούλιο είναι στην αναμονή, στη φάση αναμονής για τη συμφωνία και στα νησιά Σαλομών έχει ε, ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της κοινή γνωμοδότησης. Το Συμβούλιο είναι σε αναμονή ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της για την προσωρινή εφαρμογή. Όπως βλέπετε λοιπόν μιλάμε για ένα εξάμεινο γεμάτο προκλήσεις ε, στο οποίο ελπίζω να μπορέσω να συνεργαστώ μαζί σας ε, σε στενό συντονισμό. Το είπα και στην αρχή της περίμβασής μου, το είπε και η Πρόεδρος, η νέα συνθήκη απαιτεί από μας να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε όσο το δυνατόν πιο στεναρά και πιο υπεύθυνα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία σκέψη για την κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση της αλληλευτικής προσπάθειας. Τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τα οποία θα πρέπει να ε, ανταποκριθούμε δεν θα πρέπει να μας ε, κάνουν να ξεχνάμε τον πόσο σημαντικό ρόλο έχουμε. Η μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να διασφαλίζει μια βιώσιμη αλληλεία αλλά και αξιοπρεπές εισόδημα για τους αλληλείς, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας τους και βοηθώντας τους να, ε, καθο, να έχουν ε, πληθυσμό στις ε, παράκτες περιοχές. Αυτό θα βοηθήσει να έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία και μια πιο αλληλέγγυα Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Καλώς ορίσατε. Καλή τύχη για τις εργασίες σας κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Όπως και εσείς μόλις είπατε, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και ελπίζω μέσα από όλα αυτά τα πράγματα να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε κάποια. Η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες εδώ στην Επιτροπή μας αφορά, ε, από ό,τι άκουσα είστε ενήμερε, την ε, έγκριση της Νέας Πράσινης Βίβλου ε, και όλη την αλληλευτική κοινοτική πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας ανησυχούν, κάποιες φορές είναι αμφίβολα και απογοητευτικά. Και αυτό είναι οι σχέσεις με τις Χώρε με τις οποίες έχουμε κοινά σύνορα αλλά δεν αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτές διαπιστώνουμε κάποιες δυσκολίες διότι οι αλληλεί μα πάντα σέβονται ε, τους, κανόνες, ή όταν δεν τους σέβονται εμείς είμαστε έτοιμοι να τους επιβάλλουμε κυρώσει. Θα ήθελα να ξέρω αν κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία μπορούμε να έχουμε κάποια παρέμβαση έναντι αυτών των χωρών ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να έχει σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ αλλιέων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτών εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεων που ορισμένε φορές αλλιεύουν εις βάρος των δικών μας αλλιέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ήρθατε εδώ και μας παρουσιαστήκατε. Ε, ε, ε, έχω σύντομες ερωτήσεις. Είσαστε και υπεύθυνοι για το περιβάλλον, οπότε φαντάζομαι ότι το θέμα της ολοκληρωμένης πολιτικής των θαλασσών είναι ένα θέμα που θα σας απασχολήσει στο χαρτοφυλάκιό σας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πόσο θα ληφθεί υπόψη η αλληλεία στην ολοκληρωμένη πολιτική των θαλασσών και δεύτερον ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την κοινωνική πτυχή της ζωής των ε, ψαράδων συμφωνώ πλήρως μαζί σας διότι έχουμε ε, υπερβολικά υψηλό αριθμό ξένων αλλιευτικών στόλων στη δικά μας ύδατα και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το μέγεθος του στόλου στο τέλος. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό. Ε, εχθές το απόγευμα ήταν εδώ ο υπεύθυνος του Γραφείου Ελέγχου Αλίας στο Βίγκο και μας είπε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος έλεγχος. Αυτό λοιπόν που είναι δύσκολο να κατανοήσουμε είναι ότι δεν υπήρξε καμία μνήα εκείνη τη στιγμή και δεν υπήρξε καμία απόφαση η οποία ελήφθη σχετικά με ε, μία ομοιομορφία των προστήμων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μία λογική συνέχεια σε αυτό που συζητάμε. Πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι έλεγχοι και στη συνέχεια να υπάρχουν και ενιαία πρόστιμα. Ε, χρησιμοποιώντας όμως τα λόγια που ανέφερε ο Γενικός Διευθυντών είχε πει ότι ε, είναι ανοιχτό το πεδίο ακόμη και εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι μιας χώρας εναντίον της άλλης. Ξέρω ότι ίσως δεν είναι αυτή η πρώτη σας προτεραιότητα, είναι απλούστατα ένα θεματάκι το οποίο θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη υπόψη για να είσαστε σίγουροι για το τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Διότι το πρόβλημα προκύπτει σε ορισμένα κράτη και όχι σε άλλα. Δηλαδή υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα όπως η δικιά μου παραδείγματο χάρη όπου για ένα μικρό παράπτωμα είστε ήδη εγκληματίας ενώ σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά καθαρά. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ε, υπήρχε μία δυσκολία τελευταίως ε, σχετικά με την αλληλεία ορισμένων ψαριών και ε, ένας αλλιές χρειάστηκε να, να και οι αλλοίς τότε είχαν προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία μακροπρόθεσμη στρατηγική και να είμαστε ε, σίγουροι ότι όλοι θα θα χρησιμοποιούν τους ίδιους κανόνες και θα υπάρχει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο διότι οι υπεύθυνοι χρησιμοποιούν ένα σύστημα που υπάρχει εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια και νομίζω ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Ε, μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Κύριε Πρόεδρε, ε, καλημέρα σας. Ε, ε, εύχομαι κάθε επιτυχία στην Πρόεδρο κατά την διάρκεια της Προεδρίας της, στην Υπουργό για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα να ξέρω τι πρόκειται να κάνετε σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, διότι στην πολιτική αλληλεία θα ήθελα να ξέρω πώς αντιλαμβάνεστε και πώς προσεγγίζετε την περιφερειακή αντιμετώπιση αντιμετώπιση. Θα αναπτύξετε μία σχετική διαδικασία περαιτέρω και στην περίπτωση αυτή πώς ε, σκέφτεστε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η περιφερειακή κατανομή και όσον αφορά τη σήμανση και την οργάνωση της αγοράς αναφερθήκατε μόνο στους εσωτερικούς ελέγχους της αλληλείας θα ήθελα όμως να ξέρω ε, ποια είναι η αντιμετώπιση σας σχετικά με τις εισαγωγές λοιπόν. πολιτικές ομάδες δεν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο στους τονιστές, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει στους τονιστές και θα κλείσω έτσι το κατάλογο των αγορητών. Να σας ρωτήσω γράψιμο πως κάποιον δεν ξέρω. Andrés Barea, Sánchez Precedos, Capula Santos, Valesa, Mato Adrover, Levain y Con esto se cierra la lista. Señora Ministra... Κύριε Υπουργέ, έχετε τώρα το λόγο. Πάντω να σα πω όλα όσα γίνονται και να είστε ενημερωμένοι όλοι. Να μπορείτε όλοι να είστε ενημερωμένοι. Σε πραγματικό χρόνο. θάλασσα και τα όρια λοιπόν ηλεκτρικών περιοχών. Επίση, Επίσης έχει συλλογιστεί και κάποια επιτροπή αλίας. και ασχολείται πέραν από τα ύδατα κοντά στην Ιταλία και με άλλα και με άλλες περιοχές οπότε προωθήθηκαν λύσεις για θέματα που πάνε και άλλες θάλασσες. Δεν έχουμε αυτές τις συνήθεις προσκευές. Πάντως, αν ακόμα θεωρείτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο, με συνθήκη που έχει οριοθετήσει, με κάποιους κανόνες του παιχνιδιού, φυσικά. Και μπορείτε να απευθυνθείτε σε ποια ευλαρμόδια επιτροπή έχει συγκροτηθεί και υπάρχει. Κυρία Ρόντχορστ. Ρώτησε τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει όσον αφορά μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα. Και εδώ θα πρέπει να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Να πάμε λίγο πίσω λοιπόν όταν είχαμε λιγότερα κρατημένη. και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι εκείνη την εποχή η εικόνα των πλειοκτητών ή των ε, αλλιέων στην Ευρώπη ε, ήταν η εικόνα της εκμετάλλευσης των ε, αληθικών πόρων και καθημερινά είχαμε διάφορα συμβάντα δυσάρεστα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ελευτικά. Επιτέλεσε έργο το κοινοβουλίο σας και η Επιτροπή Γεωργίας και διάφορες προεδρίες οπότε και έγινε μια ολόκληρη πορεία που χαρακτήκε έτσι οπότε και τελικά πέρασε το μήνυμα στον ελευθερικό τομέα όσον αφορά την βιώσιμη αλληλεία. Βέβαια είναι θέμα κατά πόσον έχει αφομοιωθεί η έννοια αυτή, αλλά πάντως έχουν χωνέψει νομίζω οι Ελλήνες ότι δεν ισχύει η λογική του δόση μην σήμερα. Και ο κλάδος τώρα είναι ίσως ο πιο φανατικός υποστηρικτής της νομοθεσίας κατά της λαθραλίευσης. Οπότε και κάποια στιγμή, επί τη βάση των ε, επιστημονικών εκθέσεων και μελετών, έχουμε και τα σχέδια ανάκτησης. Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει τους ψαρότοπους να τους ε, φροντίσουμε, να τους προστατεύσουμε και να έχουμε κάποιο είδους ε, προγράμματα διαχείρισης επί τη βάση των επιστημονικών των εκθέσεων και μελετών. Να μην έχουμε εξαφάνιση ειδών, να υπάρχει κάποιο feedback ούτω ώστε να έχουμε και απασχόληση και κανονικά εισοδήματα για τους αλλίες. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ πρόσφατα. Η αλλαγή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε τώρα για βιωσιμότητα. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο είναι ευρύτερο. Μιλάμε για σεβασμό για το περιβάλλον. Και είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να καλύψει η μεταρρύθμιση της κοινή ε, αλληλευθύγης πολιτικής. Κάτι το οποίο αναμφίβολα θα είναι ένα πάρα πολύ καινοτόμο στοιχείο το οποίο πρόκειται εμείς να ε, ε, προωθήσουμε πέραν των άλλων που γνωρίζετε Αλλά να μην θεωρηθεί ότι είναι η αλληλεία μια συνεχής διαδικασία εκμετάλλευση του περιβάλλοντος είναι, είναι μια διαδικασία που εκμεταλλεύεται αλλά και υποστηρίζει το βιώσιμο περιβάλλον. Έχουμε και άλλε δραστηριότητε που θα πρέπει επίση να ληφθούν υπόψη και να υπάρχει μια ενιαία σφαιρική πολιτική. Ακριβώ όπω ε, απέκτησε την ε, σημερινή του υπευθυνότητα ο ελληνικό κλάδο, Ακριβώ όπω είναι και στην υπόθεση τη ε, προστασία του περιβάλλοντο, θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να προσέξουμε να μην ενοχοποιούμε τον κλάδο αυτόν για το ότι πάει στραβά. Γιατί υπάρχουν και άλλε δραστηριότητε και άλλοι κλάδοι που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά που εμπλέκονται εκεί. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να δούμε τι θα κάνουμε για την αύξηση της θερμοκρασίας του ύδατος, τι θα γίνεται όσον αφορά τις ε, άμεσες επιδράσεις στην αλλαγή του κλίματος και της βιοποικιλότητας στη θάλασσα και επομένως έτσι να δούμε πώς θα αποφύγουμε να έχουμε προβλήματα ελληνικών πόρων. Και να λειτουργεί και αυτόν τον τρόπο έβρεθμα αυτός ο κύκλος ε, οπότε, στον οποίο οι Ελλήνες παράγουν πάρα πολύ σημαντικός και να είναι πρότυπο προς μίμηση για άλλες δραστηριότητες. Άρα, εδώ μπαίνει το θέμα της ε, ολοκληρωμένης πολιτικής για τη θάλασσα. Φυσικά είναι και θέματα εδώ που είναι δικής μορδιότητας όπως οι θαλάσσιες μεταφορές. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ελεκτικούς πόρους και μπορούμε εδώ να αναφερθούμε στο πώς θα έχουμε σταθερότητα στη δημιουργία απασχόλησης, να έχουμε κάποια πρόγραμματα διαχείρισης απασχόληση μέσω μακροπρόθεσμα, διατήρηση και υποστήριξη του εισόδηματος, και της ε, οικονομικής δραστηριότητας. Ο κύριος ε, Γκάλερ νομίζω μας ρώτησε για διαφορετικά ζητήματα ε, όπως του κάποιους ελέγχους όπως επιβολή κάποιων οικονομικών κυρώσεων, προστήμων που επισύρουν κάποιες παραβάσεις. Όσον αφορά τους ελέγχους, ναι, έχουμε κάτι το οποίο ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία της Αλίας. Είναι ενωτικό στοιχείο, όπως είπε. είναι μια πλατφόρμα από όπου, βασίζονται και οι επιθεωρήσεις και όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Τώρα, εάν εννοούσατε άλλου είδου ελέγχους που θα μπορούσαν να προχωρήσουν παραπέρα από αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο, μήπως εννοείται και, και τις τις επαφές, τις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ε, σας θυμίζω ότι κάθε ελεύθερη συμφωνία με τρίτη χώρα προβλέπει μηχανισμούς ελεγκτικούς ούτως ώστε να τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Τόσο αφορά τα πρόστιμα. Αυτό συζητήθηκε εκτενώς στο Συμβουλίο Ελίας. Και είπαμε ότι θα πρέπει σε όλα τα να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση Από την άλλη μεριά ελέγχθη ότι θα πρέπει να ισχύσει και κατά κάποιο τρόπο η ασχή της επικουρικότητας. Είμαι ανοιχτή σε συζήτηση. Κανένα πρόβλημα να το κουβεντιάσουμε παραπέρα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αληθική δραστηριότητα δεν γίνεται πάντοτε στα πάρα πολύ κοντινά είδατα μιας χώρας γιατί μπορεί να έχουμε ένα σκάφος σκάφος χώρας που να ασκεί δραστηριότητά του σε κοινωτικά ύδατα αλλά σε άλλη χώρα μέλος. Επομένως, θα πρέπει και το θέμα των κυρώσεων να αντιμετωπιστεί ανάλογα με αυτή τη διάσταση της αληφτικής ε, δραστηριότητας. Σας ξαναλέω όμως είμαι ανοιχτή και δεν έχω κανένα πρόβλημα να ανοίξουμε το θέμα για να το συζητήσουμε. Πάντως σας επαναλαμβάνω ότι προκάλεσε συγκρούσεις απόψεων ε, το θέμα αυτό στο Συμβουλίο Ελίας. Επίσης, είχαμε και τη συζήτηση για τον Βακαλάο στο Συμβούλιο και είπαμε για τα αποθέματα. Είπαμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Είπαμε ότι θέλουμε βιώσιμη αλία στην Ευρώπη. Και μόλις έχουμε στα χέρια μας κάποιες επιστημονικές εκθέσεις, τότε θα ξεκινήσει η συνολική ε, διαδικασία με το Κοινοβούλιο, με, το, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να τρέχουμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια μεγαλύτερη και πιο μακροπρόθεσμη σταθερότητα στα αποθέματα. Κάτι άλλο τώρα το οποίο ανέκυψε ήταν η περιφερειοποίηση, κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Γκρόμπετσικ. Ε, προσοχή εδώ πέρα, μην γίνεται σύγχυση. Γιατί έχουμε την ε, περιφερειοποίηση, η οποία πολλές φορές μπερδεύεται με την επανεθνικοποίηση. Όχι, δεν θέλουμε εμείς ως Προεδρία την επανεθνικοποίηση. Γιατί έτσι θα είχαμε την ταφόπετρα στην κοινωνική πολιτική. Και όσον αφορά την περιφερειοποίηση, πρέπει να διακρίνουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή η ζώνη στην Ευρώπη ή σε κάποια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα. Και έχουμε κάποια σαφή παραδείγματα για θέματα που έχουν ανακύψει. Έχουμε α πούμε την απότερη περιφέρεια και τι σχετικέ περιφερειέ τη κοινότητα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για συγκεκριμένε περιοχέ και αυτό δεν αφορά μόνο την ελευτική πολιτική αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια ούτω ώστε να έχουμε μια κοινή ελευθερική πολιτική αλλά και να μπορούμε να είμαστε σε θέση εδώ να καλύψουμε όλες τις διαφορές που αποτελούν τον πλούτο μας μια που έχουμε τέτοια ποικιλία και πολυμορφία στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε ή να αξιοποιήσουμε μέσα από την η ελληνική πολιτική. Βεβαίω και πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί. Βεβαίω και θα πρέπει αυτό να του αφορά όλου και θα πρέπει σε αυτήν την προσπάθεια να είμαστε ενωμένοι. Έτσι θα βλέπω εγώ τα πράγματα. Να αναδείξουμε την ε, πολυμορφία μας και να την σεβαστούμε. Και σας επαναλαμβάνω ότι για μένα με τίποτα θα πρέπει αυτό να μας οδηγήσει σε πανεθνικοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στίβενσον, σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Υπουργό ε, για τη σημερινή μας συνάντηση. Έχω δύο ερωτήσεις σχετικά με την επανεθνικοποίηση ε, δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε ε, να υπαγορεύσουμε ένα γενικό καλούπι για την ε, περιφερειοποίηση. Θα παρακαλούσα λοιπόν ε, να αφαιθεί στα κράτη, στην κρίση των κρατών μελών πώς θα διατυπώσουν προτάσεις για τις συγκεκριμένες ε, περιφέρειες Βεβαίως ε, υπό την εποπτεία και την τελική ευθύνη του Συμβουλίου, της Επιτροπής και βεβαίως και του Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά ε, τα αποθέματα είτε τη χάνουν υπερβολικής εκμετάλλευση στην Ευρώπη ή έχουν καταρρεύσει. Ε, θα χρηματοδοτήσουμε μη έναν εξυγχρονισμό του αλληλευτικού μας στόλου για να μπορέσει μπορέσει ο τομέας να παραμείνει βιώσιμος ε, αντί ε, να ε, χρηματοδοτούμε γιατί όμως να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα έτσι όταν υπάρχει υπερβολική εκμετάλλευση της αλληλείας γιατί να χρηματοδοτήσουμε τον αλληλευτικό στόλο. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ κυρία ε, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ σαν εκπρόσωπο της Ισπανικής κυβερνήσεως ε, που ήρθατε εδώ και πιστεύω το θέμα μας ακόμη εκρεμεί. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της ε, Ισπανικής Προεδρίας για την εφαρμογή των ε, μεταφερομένων ε, προσωπικών ποσοστώσεων. Βλέπω την ε, Προέδρο κυρία Φράγκα που χαμογελάει, εγώ όμως δεν γελάω και όπως ο κύριος Κάλαγκερ είπε προηγουμένως θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε για να υπάρχουν ε, ε, να υπάρχει σεβασμός των ποσοστώσεων στην Ευρώπη και τέλος θα είμαι σύντομος συμμερίζομαι την ανησυχία της Προέδρου μας για την ε, εγγραφή του κόκκινου η ε, ε, ε, στα θέματα που είναι επικίνδυνα. Η κυρία Αντρέ Βάιρα, ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. εχθε ξεκίνησε η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στην κοινή αλληλευτική πολιτική και θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα μορφή διαχείριση. Το θέμα τη αλληλευτική προσπάθεια, πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε δηλαδή. Θέλουμε να μας πείτε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα θέματα της διαχείρισης, σεβόμενοι και το περιβάλλον, όπως είπατε κι εσείς. <laughs> Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το 70% του πλανήτη μας είναι νερό και από αυτά το 50% τουλάχιστον είναι αλμυρό νερό, θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ίσως γυναίκα νομίζω ότι θα ταυτίζεστε απόλυτα, να ε, λάβετε υπόψη και το θέμα της ισότητας των φύλων. Στην Ισπανία το θέμα αυτό είναι προτεραιότητα. Είμαστε σε προεξάρχοντα ρόλο επί του θέματος. Τι, πώς θα ενθουσιαστώσετε λοιπόν και τη συνιστόσα του φύλου στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ώστε οι γυναίκες να έχουν και το πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχουν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε και το ίμιση των αλλιών. Ευχαριστώ κύριο Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλωσορίσατε κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να μπορέσετε εσείς να ξεπεράσετε αυτό τον κοινοβουλευτικό μαραθένιο τον οποίο έχετε ξεκινήσετε ε, που έχετε εμφανιστεί ως προεδρεύουσα σε διάφορες επιτροπές. Η προεδρία σας θα είναι ιδιαίτερο σημαντική, διότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε πολύ σημαντικές στιγμές. Νομίζω ότι εσείς ε, είστε μία από τις ε, προεδρίες που αναλαμβάνουν μετά από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε πλέον το 17 μήνο της Προεδρίας. Είστε μία από τις κοινέ Προεδρίες και ελπίζω ότι ε, θα μπορέσετε να συνδράμετε ώστε η αλληλεία να θεωρηθεί ε, πρωταρχικός παράγοντας και οι αλληλείς να λάβουν το ρόλο που τους αρμόζει. Πρώτον, ε, μιλάμε για μια κοινή αλληλευτική πολιτική που πρέπει να μεταρρυθμιστεί, που θα λάβει υπόψη της και τους πόρους και εσείς μιλήσατε για κοινέ ε, αγορές αλληλείας. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό και επίσης θα ήθελα να μου πείτε, ε, είπατε κάποια πράγματα για την ε, προγράμματα διαχείριση Γαύρου, Σαυρουδίου και Βακαλαίου του Ατλαντικού. Θα ήθελα κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες. Ευχαριστώ και τέλο, για το τέλο του δεύτερου γύρου, ο κύριο Καπούλα Σάντο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, κύριε Υπουργό, να τη ευχηθώ. Σας γνωρίζω και γνωρίζω ε, και τις πολιτικές σας ικανότητες, αλλά ε, και γνωρίζω ότι η Ισπανία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είστε και υπουργό Περιβάλλοντος ταυτόχρονα, γεγονός που αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα αν μιλάμε για την αλληλεία. Κάποιοι συνάδελφοι το είπαν, ε, θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάποια πράγματα για το μέλλον της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Το πιο ευαίσθητο σημείο είναι το θέμα της διαχείρισης των πόρων. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπει η Προεδρία το θέμα των μέσων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ε, ποια θα πρέπει να κυρωθούν, ποια θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν, ποια θα πρέπει να επανεξεταστούν για να μπορούμε να δούμε πώς θα έχουμε βιώσιμους πόρους. Ευχαριστώ, Υπουργό, για να απαντήσει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της επανεθνικοποίησης που έθεσε ο κύριος Στίβενσον. Νομίζω ότι η πρώτη μου απάντηση ήταν μια απόπειρα να σας πω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όμως δεν θα πρέπει να φτάνουμε στα άκρα. Εγώ μιλούσα για μια κατάσταση στην οποία δεν ισχύει να έχουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική αν δεν γίνεται διαφοροποίηση ε, λόγω περιφερειακής συνιστώσεως, λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ε, και να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και η επανεθνικοποίηση κατά την άποψή μας θα ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Θα ήταν σαν να εξατομικεύουμε τα πάντα και θα είχαμε μια αλληλευτική πολιτική ε, που θα είχε μια ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, ανά χιλιόμετρο των ακτών μας. Το μόνο που θα μας έδινε θα ήταν κάποιοι περιορισμοί και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλοι για την κοινή ελευτική πολιτική. Αυτό που δεν θα ήθελα είναι να παρερμηνεύσετε ε, αυτό που σας είπα. Ναι, μεν κοινή αλληλευτική πολιτική, με ένα πολύ μεγάλο ναι, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε χώρας και κάθε περιοχής θα λαμβάνονται υπόψη, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να βάζουμε ονοματοπώνυμο σε κάθε αλία και σε κάθε σκάφος, διότι κατόπιν θα μιλάμε για ένα ατομικό σύνολο συμφερόντων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Επιπλέον, ναι μεν είπα ότι υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία λαμβάνουμε υπόψη ε, από το παρελθόν, αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είπα στην πρώτη παρέμβασή μου, αλλά αν θυμάμαι καλά, αυτό, αυτή η έννοια εισήχθη το 2002 και τότε ήταν η περίοδος στην οποία ετέθησαν οι βάσεις για τα περιφερειακά συμβουλευτικά ε, για τις περιφερειακές ενός αλληλείας, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν εξαπλωθεί και καλύπτουν ε, και τα συγκεκριμένα είδη αλληλείας και τη συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία που εμφανίζουν κάποιοι συγκεκριμένοι αλληλευτικοί τομείς και τα συμφέροντα των αλλιέων. Η βελτίωση αυτών των μέσων και η δημιουργία παρόμοιων μέσων θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι, και αυτό το παρουσιάζω και ως ιδέα για τη συζήτησή σας, ε, μια κατάλληλη άγουσα για να επιτύχουμε αυτό το οποίο θέτετε εσείς. Υπάρχουν και θέματα ανάγκης ή μη ανάγκης κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ε, εκεί νομίζω ότι ήμουν σαφής. Σας είπα και ένα τεράστιο ναι και θεωρούμε ότι και ιστορικός ήταν ένα από τα κοινά πολιτικά θέματα που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πάροδο των ετών μιλάμε για περισσότερες κοινέ πολιτικές, αλλά ιστορικώς η αλληλεία ήταν αυτή που ήταν η πρώτη κοινή μας πολιτική. Όταν γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε ένας πάρα πολύ σαφός, σαφής λόγος για τη γέννησή της. Αν το είχε τότε λοιπόν, σήμερα το έχει περισσότερο από ποτέ. Και αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Γιατί πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τον εξυγχρονισμό. Δεν θα πρέπει εδώ να χρησιμοποιούμε λανθασμένη έννοια, διότι ο εξυγχρονισμός δεν σημαίνει απαραίτητο μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Να θέσω κι εγώ μια ερώτηση και τη θέτω για να μείνει ως ρητορικό ερώτημα. Δεν θεωρείτε ότι οι Ευρωπαίοι αλλιές έχουν δικαίωμα να ζουν και να διεξάγουν την εργασία τους σε καλύτερες συνθήκες από ό,τι πριν από κάποια χρόνια. Οποιοδήποτε ε, επάγγελμα προωθείται σε θέματα ασφάλειας, ε, ε, σε θέματα ε, καλύτερου εισοδήματος, γιατί να μην προχωρήσει και το τομέας της Αλλίας. Και επιτρέψτε μου τώρα ως καταναλωτής να σας μιλήσω. Εγώ ως καταναλωτής απαιτώ όλο ένα και περισσότερη ασφάλεια σε ό,τι επιλέγω. Αν επιζητώ λοιπόν την ε, ασφάλεια σε ένα ε, ε εργοστάσιο που παράγει ε, τρόφιμα γεμιστά. Θα πρέπει να τους δίνεται για παράδειγμα η συνδρομή για όλα τον εξυγχρονισμό. Υπάρχει επιδότηση για τον εξυγχρονισμό. Αν μιλάμε για την αλληλεία, τα σκάφη είναι το, ο αντίστοιχος εξυγχρονισμός που σας μιλούσα για τον εξυγχρονισμό των ε, εργοστασίων. θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα παραδείγματα, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να μιλάμε και για πολύ περισσότερα θέματα. Μας θέσατε παράδειγμα τα φορτηγά οχήματα. Υπάρχουν πολλά σχέδια. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικά σχέδια για ε, ανανέωση του στόλου των φορτηγών οχημάτων. Το θέμα της ασφάλειας τίθεται και από πλευράς περιβάλλοντος. Θέλουμε για τα φορτηγά οχήματα να έχουμε ένα πιο σύγχρονο στόλο, ένα πιο σύγχρονο ε, ε, αποθεματικό που θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα θα πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και να σκεφτούμε ότι ναι μεν υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν επιδοτήσεις αλλά επειδή τις λαμβάνουν υπό διαφορετικό σκεπτικό μπορεί να τραβούν περισσότερο την προσοχή μας, λιγότερο συγγνώμη την προσοχή μας. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια σύγκριση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δημιουργείται είτε μέσω είτε άμεσα ε, σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δείτε εκεί ότι θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, κάποια πράγματα που έκανα εγώ σε επίπεδο της χώρας μας πραγματικά ε, τράβηξε την προσοχή. Πρόκειται κάτι, για κάτι λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού και που θα χρησιμεύσει ίσως ώστε να υπάρχει η διαφάνεια που θέλουμε να διαβιβάσουμε και στους πολίτες Και επειδή ακριβώ βρισκόμαστε και σε αυτό το νέο στάδιο της συναπόφασης, θα μπορέσουμε ίσως να προχωρήσουμε πολλά πράγματα και να πάψει να ισχύει ο μύθος ότι η αλληλεία και η γεωργία είναι αυτοί οι οποίοι ε, κατασπαταλούν τον ε, προϋπολογισμό, είτε τον ευρωπαϊκό είτε τον ε, προϋπολογισμό των κρατών μελών. Μιλήσαμε και για τις ε, ε, ατομικές μεταφορές. Κάποιες λεπτομέρειες. Η κατανομή των ποσοστώσεων της αλληλείας θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εγγύηση προς τις επιχειρήσεις, ε, διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο μπορούν να ηλιεύσουν, αλλά εάν δεν επαρκούν, σε κάποιες περιπτώσεις έτσι συμβαίνουν με τους ευρωπαϊκούς στόλους, δεν θα επαρκούν για το εισόδημά τους. Τα υφιστάμενα συστήματα μέχρι τώρα τα υπόλοιπα λαμβάνονται υπόψη μόνο εντός ε, κάθε κράτους μέλους. Εάν υπάρχει αύξηση μιας επιχείρησης, αυτό θα γίνεται εις βάρος άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κράτους μέλους. Αυτό είναι εθνική πολιτική. Δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική αν θέλουμε να σκεφτούμε το σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφού δεν υπάρχουν πλέον σύνορα, ε, θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι ιδέες τις οποίες θα ήθελα να σας διαβιβάσω, ώστε να γίνει αυτή η ανοιχτή συζήτηση και να ε, καταλήξουμε ίσως σε κάποια αποτελέσματα. Υπάρχουν βέβαια και δυσκολίες. Θα μπορούσε τα πράγματα να πάνε πολύ καλά όταν μιλάμε για επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους. Αν όμως ε, μιλάμε για τον ε, στόλο των ε, μικροαλλιέων και εδώ να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων αλλιέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι όλα τα ωφέλη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε, άλλους, ε, σε άλλες επιχειρήσεις. Όπως μιλήσαμε για περιφερειοποίηση εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και ένα μέσο το οποίο θα στοχεύει στην τελειότητα βάσει και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα θα βοηθήσει και τη βιωσιμότητα του στόλου που έχουμε στην Ευρώπη. Κατά την άποψή μας ε, είναι πολύ λογικό, αλλά κατά την άποψη κάποιων άλλων είναι ένα μέσο το οποίο είναι επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση. Κατά την άποψή μου ναι ότι θα χρειαστούμε περισσότερη προσπάθεια και θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όντως ισχύει. Αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε και σας προσφέρω τη συνεργασία μου. Να περάσω τώρα σε αυτά που ρώτησε η κυρία Αντρέ Βαρέα για την ανθρώπινη διάσταση και την ισότητα των φύλων. Εχθές ε, πήγα και στην Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου και μίλησα για την ανάγκη ισότητας στον αγροτικό κόσμο. Όταν μίλησα για ισότητα στον αγροτικό κόσμο δεν αναφερόμουν φυσικά μόνο στις γεωργικές δραστηριότητες ε, ή στι κτηνοτροφικές δραστηριότητες που μπορεί να έχουν κάποια άμεση σχέση επί του θέματο, αλλά ε, και ισότητα στις αλληλευτικές δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, στο παρελθόν δεν είχε συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επειδή όμως είναι κάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη της υπαίθρου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την αλληλεία Πριν από κάποια χρόνια όταν μιλούσαμε για ε, γεωργικές επιδοτήσεις ε, στο IFOP, ε, κάναμε μία διάκριση μεταξύ αυτών που κάνουν μία γενή δραστηριότητα αλληλείας και γεωργίας και των νέων. Δεν έγινε όμως κάτι συγκεκριμένο για τις γυναίκες. Αν λοιπόν ο καθένας από μας ε, δει τον αλλιευτικό τομέα στη χώρα του, θα διαπιστώσετε ότι οι γυναίκες σε κάθε μία από τις χώρες σας, στον τομέα της αλληλείας, κάνουν πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες. δραστηριότητες πολύ συγκεκριμένε που ε, παρόλα αυτά δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη. Μιλάμε για επισκευή δικτυών. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε επίσης και για ε, ε, δραστηριότητες στην αλία θαλασσινών ή την πρώτη επεξεργασία ψαριών. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συζήτηση που θα γίνει για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτικής, να δώσουμε μια νέα όθηση και να εκμεταλλευτούμε και το νέο πλαίσιο διαρθρωτικών επιδοτήσεων στην Αλία και στα μελλοντικά μέτρα στήριξη τη παράκτεια αρίας, διότι κυρίω μιλάμε για παράκτε δραστηριότητε, να προσπαθήσουμε να λάβουμε περισσότερο το ρόλο τη γυναίκε για να δοθεί και ιδέουσα σταθερότητα στην οικογενειακή οικονομία σε πολλές περιοχές οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από την αλία. Υπάρχουν επίσης σύλλογοι οι οποίοι ουσιαστικά εξαρτώνται από την ε, Ευρωπαϊκή Διαρθρωτική Πολιτική και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε μεταξύ μας και να υπάρξει η ισότητα που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο της αλληλείας ώστε να μην διαφοροποιείται από κανέναν άλλον τομέα. Κάποιες χώρες, κάποια κράτη-μέλη το έχουν ήδη κάνει ή το έχουμε ήδη κάνει. Αλλά κυρίως χρειαζόμαστε και αυτή την ε, ευρωπαϊκή σκέπη η οποία θα δώσει μια πιο μεγάλη ανθρώπινη διάσταση. Ο κύριος ε, Σάνσες Πρεσέδο είπε ότι θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Δεν ξέρω αν ε, ε, θα τα καταφέρω. Πραγματικά όντως ήρθα σε τρεις επιτροπές αυτή την εβδομάδα και ήμουνα και την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, Ολομέλεια, οπότε μπορεί και να είναι ρεκόρ εμφανίσεων, αλλά νομίζω ότι ε, όλα αυτά τα πράγματα είναι πέρα από μία απλή νομοθεσία, έναν απλό κανονισμό. Πάντα η συζήτηση, ο διάλογος μπορεί να αποφέρει καρπούς και πάντα μπορούμε να συνεισφέρουμε ένα λιθαράκι παραπάνω για να ε, υιοθετήσουμε και τα κατάλληλα μέτρα σε αυτή την περίπτωση ε, ε, για την αλληλεία που να είναι και τα καλύτερα δυνατά. Μιλήσατε και για την κοινή οργάνωση αγοράς και για τα προγράμματα διαχείρισης ε, του ΓΑΒΡΟΥ, του Σαβριδίου και του Βακαλάου του Ατλαντικού. Στο θέμα της κοινή οργάνωσης αγοράς, ε, ξέρουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για μια νέα κοινή οργάνωση αγοράς. Αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλωσε και πλέον δεν προσαρμόζεται στις ε, πραγματικές μας ανάγκες. Και θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση τόσο για τις ελευτικές δραστηριότητες όσο και για την ηχθοκαλλιέργεια. Και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαφοροποίησεις. Τα τελευταία χρόνια οι εισαγωγές αλληλείας ε, όλο αυξάνονται και όταν ε, ξεκίνησε αυτή η κοινή οργάνωση αγοράς δεν υπήρχε ούτε το ειδικό βάρος ούτε οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν ε, σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να πρικοδοτήσουμε και την κοινή οργάνωση αγοράς Δεν ε, θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση να δεν μιλάω για καταστρατήγηση του ελεύθερου εμπορίου, μιλάμε για αμοιβαιότητα και μιλάμε και για διασφάλιση πληροφοριών και εγγυήσεις προς τους καταναλωτές σε κάποιες περιπτώσεις με μέσα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα όπως η οικολογική επισήμανση την οποία ανέφερα και σήμερα. Όσον αφορά τώρα στο Γαύρο, συγγνώμη, στο Βακαλάο του Ατλαντικού, να σας πω ότι είμαστε σε κατάσταση αναμονής, περιμένουμε την επιστημονική γνωμοδότηση και όταν θα λάβουμε την επιστημονική γνωμοδότηση θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε και το σχέδιο. Για το Σαβρίδι, θα μπορούσε ίσως να γίνει η πρώτη κοινή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, νομίζω ότι υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις και θα αναζητήσουμε ημερομηνίε για να γίνουν ε, τριμερείς συνεδριάσεις και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, και να λύσουμε μικροδιαφορές κατά την άποψή μου. για το γάβρο τώρα πρόκειται για ένα είδος που ναι μεν δεν αφορά όλο τον ευρωπαϊκό στόλο αλλά είναι πολύ σημαντικό για το γαλλικό ή τον ισπανικό στόλο και επομένως ε, η έγκριση του σχεδίου θα μπορέσει να μας επιτρέψει να ε, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια εκμετάλλευσης για ένα απόθεμα με το οποίο αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Χρειάστηκε να κλείσει η ζώνη αλίευσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά και για κάθε κράτος μέλος που είχε στόλο που έκανε αλία γάβρου έγιναν τεράστιες επιστημονικές προσπάθειες για να γνωρίζουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ε, από δύο ε, έρευνες που έγιναν ε, κάθε χρόνο και κάθε χρόνο είχαμε όλο και περισσότερους εμπειρογνώμονες για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις για την διάσωση του αποθέματος. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό την ισορροπία της βιωσιμότητας, την οποία ε, ζήτησε και ο ίδιος ο κλάδος ε, μέσω του Περιφερειακού Συμβουλευτικού Οργάνου των ε, Δυτικών Υδάτων. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι στο παρελθόν δεν το καταφέραμε. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερη αβεβαιότητα, διότι επειδή μιλάμε για ένα μικρό στόλο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις που υπάρχουν και για τις ε, επιχειρήσεις μεταποίησης. Τέλος, ο κύριος Καπούλας Σάντος ανέφερε όλα τα θέματα βιωσιμότητας εν γέννη. Σας είπα στην πρώτη μου παρέμβαση κάποια πράγματα για τη βιωσιμότητα για να ολοκληρώσω λίγο τις πληροφορίες που σας έδωσα, θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούμε για τους παρόντες στόχους της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και ο βασικός στόχος είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων μας για να υπάρχουν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα επιτρέψουν στους αλληλείς να ζουν από αυτή τη δραστηριότητα και να μπορούν να ζουν στο μέλλον από αυτή τη δραστηριότητα πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή η τριπλή συνιστόσα, η κοινωνική, η οικονομική και η περιβαλλοντική, ορισμένες φορές είναι δύσκολο να την εξηγήσουμε και κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι και δύσκολη στην εφαρμογή της. Εγώ θα ήθελα όμως να το δείτε λίγο αντίστροφα το ζήτημα. Εάν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε κάτι από πλευράς περιβάλλοντος ή ε, δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε με βιώσιμο τρόπο, δεν θα έχουμε αποθέματα. Και αν δεν έχουμε αποθέματα, δεν θα έχουμε ούτε οικονομικό πλούτο, ούτε κοινωνικό πλούτο. Επομένως, δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως δυσκολία, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να διατηρηθεί ο πλούτος μας βάσει αυτών των τριών στόχων. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και ας δούμε απλώς τι σημαίνει ένα πρόγραμμα ανάκτησης ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης. Τι σημαίνει ένα σχέδιο πρόληψης στην αλία. Σημαίνει να προλάβουμε καταστάσεις ε, ε, που μπορεί να μας οδηγήσουν στην κατάρρευση. Ε, ορισμένες φορές το τοπίο ήταν τελείως διαφορετικό. Θέλουμε λοιπόν να τελειοποιήσουμε, να έχουμε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που θα τις χρησιμοποιούμε ως βάση και από εκεί και πέρα να λαμβάνουμε συνειδητές αποφάσεις που θα μας δώσουν την ασφάλεια που θέλουμε για το μέλλον. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Άλλοι τέσσερις θέλαμε λόγο για να ολοκληρώσουμε. Πρώτος ο κύριος Βαλέτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία, κυρία Υπουργέ. Από αυτά τα οποία μας είπατε ε, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η ε, Προεδρία της Ισπανίας ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει αντί να αποκεντρώσει το οποίο έχει και καλά και κακά στοιχεία οπότε θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με το κοινοτικό σύστημα ελέγχου τα τελευταία χρόνια όπου διαπιστώνουμε μία όλο και μεγαλύτερη παρεμβολή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, στα θέματα της αλληλείας γλυκών κουνέρου. νερού ε, θα χρειαζόταν λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία και ε, να υπάρξει ε, ένα ε, σύστημα ελέγχων το οποίο θα εξετάζει το θέμα της υδατοκαλλιέργειας και των καλλιεργειών των εσωτερικών υδάτων γλυκού νερού δηλαδή όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κόστος προσαρμογής διαφορετικών τομέων, διαφορετικών οικονομικών συστημάτων και άλλων παραγόντων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιστεύω ότι κατόπιν αυτού ότι πρέπει να απορρίψουμε αυτή την πολιτική. Εσείς όμως τι πιστεύετε. Μάτω. Πριν από λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να πω την ε, υποψήφια επίτροπο ότι η απότερη περιφέρεια έχει διομορφίες και άρα θέλει και ιδιαίτερη ε, μεταχείριση. Ε, οπότε το ξέρετε εσείς αυτό και βεβαίως έχει την ευκαιρία την υπέροχη ευκαιρία η Ισπανική Πρόεδρε από την Κύπρο να τη χάσει ούτως ώστε κάτι να κάνει για αυτές τις περιοχές. κάτι να γίνει όσον αφορά την αλλήλεια και όσον αφορά την διατοκαλλιέργεια που να ε, αντιστοιχεί στις πραγματικές ε, ανάγκες. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, παραδοσιακός ελευτικός τόλος, ούτως ώστε η παράκτεια αλλήλεια να μπορεί να έχει τη μεταχείριση την ιδιαίτερη που της αξίζει. Να είναι προτεραιότητα αυτό δηλαδή στην ε, Προεδρία. Σας παρακαλούμε λάβετε υπόψη αυτά τα αιτήματα και προχωρήστε προς λήψη αποφάσεων. Φράγα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ε, καλωσορίζω την ε, κυρία Υπουργό στην Επιτροπή μας. Ε, είχαμε ακούσει πριν από εσά τη Σουηδέζα Υπουργό σχετικά με την ρύθμιση των ελέγχων και μία μεγάλη αποτυχία του προηγουμένου έτους ήταν ε, η ρύθμιση της βορείου θαλάσσης. Μας είπατε βέβαια ότι εσείς δεν ήρθατε εδώ σαν Ισπανίδα υπουργό, αλλά σαν εκπρόσωπος της Προεδρίας. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω διότι ήξερα ότι η Ισπανία ήταν κατά της τεχνικής ρυθμίσεως ε, των ε, ε, ε, της Βορείου θαλάσσου, θαλάσσης κατά της αυξήσεως του μεγέθους των ματιών των δικτυών. Παραδείγματος χάρη εσείς τι θα πιστεύατε ότι πρέπει να γίνει εφόσον πιστεύετε ότι χρειάζεται μια κοινή αλληλευτική πολιτική για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα κοινά αποθέματα τα αλληλευτικά τα οποία έχουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μέλη έχουν συνεργαστεί σειρά ετών για την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανονισμού. Σχετικά τώρα με την ε, υπερβολική χρήση αλλιευτικού δυναμικού ε, υπάρχουν ε, μικρότερα στόλοι που έχουν παραδείγματο χάρη το μισό μέγεθος από το ισπανικό αλλά 27% περισσότερα αλλιεύματα από τα ισπανικά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να μειωθούν οι ανισότητες και μιλώντας για επιδοτήσεις η ε, κοινή αλλιευτική εξωτερική πολιτική ιδίως προωθεί τους Ισπανούς αλληλείς οι οποίοι μπορούν να ψαρέψουν αλλού. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδοτεί ε, την ε, αλληλεία εμπορία των Ισπανών σε, στα χωρικά ύδατα των ε, υποανάπτυξης χωρών. Μιλπάω. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για το όσα μας είπατε και καλή τύχη σας ευχόμαστε για τους μήνες της Προεδρίας και να έχουμε καλή συνεργασία ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, στις οποίες βρίσκεται ο κλάδος. Όσον αφορά τώρα τις ε, αληθικές συμφωνίες, σας παραπέμπω στα όσα γίνεται στον Ειδικό Ωκεανό και ε, στα, τις συνθήκες της ε, Σομαλίας και είχαμε την σχετική πειρατεία εκεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει να ανοίξουν οι καινούργιες αληθικές περιοχές ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα γιατί αλλιώς αμαυρώνεται η εικόνα του στόλου που έχει σημεία ευκαιρία ευρωπαϊκή και αλλιεύει στον Ινδικό. Πέστε μας τι μπορεί να κάνει τόσο ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του κλάδου και να μπορέσουν να κινηθούν οι αλλιείς μας δυνάμει αυτών των συμφωνιών. Πρόσφατα δίναμε ένα ψήφισμα και ζητούσαμε να καλυφθούν τα ελληνικά από την προστασία που έχουν στην επιχείρηση Ατλάντα τα εμπορικά σκάφη. Γιατί έχουμε εδώ πέρα και την ε, ανθρώπινη πτυχή. Είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν απαχθεί. Έχουμε αυτούς όλους που ζουν το οικογενειακό τους δράμα και το προσωπικό λόγω της ε, πειρατείας και των απαγωγών. Πέστε μας αν θέλετε να προωθήσετε κάποιο είδους πρωτοβουλία ούτως ώστε να καλύψετε όλους αυτούς και από οικονομικής πλευράς ούτως ώστε να μπορέσετε να καταλήξετε και σε κάποια μέτρα υποστήριξης. Τώρα για πέστε μας για την Σαρδέλα. Για το Γαβρό. Πού ε, θα πρέπει να συνεργαστείτε με, τη, με το Κοινοβούλιο. 90% για την Ισπανία, 10% για τη Γαλλία σαν ποσοστώσεις και μετά από αυτή την παραχώρηση του 20% και 100.000 τόνων ε, έγινε αυτή η παραχώρηση προς τους Γάλλους όμως προς έκπληξη δυσάρεστη των αλλίων το Συμβούλιο έδωσε άλλους 100 τόνους στους Γάλλους τι λέτε και όσον αφορά την περιφερειοποίηση για πέστε μας συμφωνείτε με άμεση συμμετοχή των περιφερειών όσον αφορά τις περιφέρειες που έχουν αληθικέ αρμοδιότητες. Ευχαριστώ λέει και δίνω το λόγο στην Υπουργό. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιέζει ο χρόνος. Οπότε θα σας τα πω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο κύριος Βαλέσα μας είπε για Νομίζω υπήρξε κάποια παρεξήγηση όσον αφορά την, την απορρίθμιση, την, την, την κεντροκατευθυνόμενη πολιτική και, και το αντίθετο. Εδώ λέμε για κοινή ελευθερική πολιτική όπου θα έχει αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία ε, του προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θέλετε να το πείτε κεντροκατευθυνόμενη ρύθμιση. Μια που μιλάμε για την Ευρώπη στο σύνολό τη, τότε συμφωνώ μαζί σα. Αν εσείς το λέτε αυτό αποκέντρωση, αν θεωρείτε ότι είναι αποκέντρωση το κάθε κράτος μέλος να εφαρμόζει διαφορετική πολιτική, τότε δεν συμφωνώ μαζί σας σε αυτή την περίπτωση. Κοίταξτε, το θέμα είναι περίπλοκο, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια κοινή πολιτική που όμως να μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες καταστάσεις. Ως πρόεδρε, εμείς αυτό που δεν συμφωνούμε είναι η κάθε χώρα να εφαρμόζει μια διαφορετική ελευθερική πολιτική μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επίσης, αυτό κολλάγει σε αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος ε, Μάτο. Και το είπα και εγώ ίδιο προηγουμένως. Για κάποια άλλη ερώτα απάντηση. Ας πούμε για την απότερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Καλή από το άρθρο 349 της Νέας Συνθήκης και νομίζω ότι η Ελία άμεσα πειράζεται λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών από αυτή τη ρύθμιση. Άρα θα πρέπει να δείξουμε την αντίστοιχη ευαισθησία όταν θέλουμε να έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες περιοχές και ζώνες στην περιφέρεια της Ένωση από όπου και προέρχεται ο κύριος Μάτο. Και υπάρχει και άλλο παράδειγμα των, της αντίστοιχης περιοχής της Πορτογαλίας. Και η Γαλλία έχει όμως τέτοιες περιοχέ από τρει περιφέρειες. Οπότε, το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι βέβαια το να δείξουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία ούτως ώστε και από δική μα πλευρά σε αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί από την ε, αυριανή κοινή ελληνική πολιτική. Ούτω ώστε οι, οι αλίες σε εκείνες τι περιοχέ να καλυφθούν σε όλες τους τις ανάγκες. μια που εκεί ο ελευθερικός τόλος είναι παράκτιας αιλίας και παραδοσιακής υφής. Επίσης, δούμε τι θα γίνει με τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται και για την ηχθειοκαλλιέργεια. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε έρευνα, έχουμε την καινοτομία σε αυτό το επίπεδο, οπότε και εκεί πέρα αναπτύσσεται η χθιοκαλλιέργεια ακριβώς γιατί υπάρχουν οι κατάλληλες ε, συνθήκες. Μην ανησυχείτε, όλα αυτά πάντοτε τα υποστηρίζαμε και αυτά τα χαρακτηριστικά αυτά εκείνων των περιοχών ε, πάντοτε τα λαμβάναμε όπως και τα προωθούσαμε. Κατόπιν μιλήσαμε για τα τεχνικά μέτρα και τη σχετική νομοθεσία. Κάτι γνώμη μου, δεν υπάρχει δισταγμός να προχωρήσουν προ τέτοια μέτρα. Απλώς ακόμα δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Προχωρήσαμε αρκετά γρήγορα και γι' αυτό και δεν σημειώθηκε απαραίτητη συνένεση μεταξύ κρατών μελών. Δεν είναι όμως ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το αντίθετο. Όλοι πιστεύουμε ότι χρειάζονται τεχνικά μέτρα αλλά δεν είχαν γίνει ακόμα οι απαραίτητες ε, συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κάτι πολιτικού χαρακτήρα είχαν γίνει. Οπότε γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται να υπάρξει μια διαδικασία και να οριμάσει κατά φυσικό τρόπο το θέμα το, το οποίο είναι κάτι το οποίο ισχύει για οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε νόμο. Επίση, μιλούσαμε και για την υπεραλίευση ή την, την, υπερβολή σε επίπεδο αληφτικού στόλου, αυτό πάντοτε θα πρέπει να αντιστοιχεί στο τι αληθικούς πόρους έχουμε. Δεν θα πρέπει να γενικεύουμε γιατί έχουμε κάποιους ε, στόλους οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι τέλεια στους, στους πόρους και σε άλλες περιπτώσεις ε, όντως έχουμε δυσαναλογία μεταξύ στόλου και πόρων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση τέτοια για να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα ή σχέδια. Για να μπορούμε να υιοθετήσουμε τα αναγκαία μέτρα και έτσι να φτάσουμε στην ευθυγαμισμένη ανάπτυξη στόλου με τους πόρους και να φτάσουμε στη βιώσιμη αλία. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τη αλίας για συγκεκριμένε περιοχέ, οπότε η κοινή αλληλεία είπαμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε χρειάζεται έναν ε, συγκεκριμένο σχεδιασμό που να προσαρμόζεται σε κάθε είδος ε, σε κάθε είδος ε, ψαριού. Ας πούμε λέμε για το γάβρο, λέμε για το σαφρίδι, ε, για το βακαλάο και αντίστοιχα προχωρούμε και εμείς για να δούμε κατά πόσο θα κάνουμε αυτή την, την αντιστοίχηση στόλου ε, πόρων. Θα πρέπει να ε, ενεργούμε παντού όμως με ενιαίο τρόπο και πάντοτε λαμβάνοντα υπόψη τους ειδικού πόρους που υπάρχουν. Κυρία Μπιλμπάου τώρα που αναφέρθηκε σε κάτι που θα πρέπει πρώτα πρώτα να το διευκρινίσω γιατί έχουμε κάποια θέματα τα οποία έθεσε και αφορούν την εθνική, ισπανική πολιτική. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί εδώ δεν παρίσταμε ως ε, υπουργό. Επομένω, δεν μπορώ να σας πω όσον αφορά τις, ε, ε, τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας και τις αρμοδιότητες τους, δηλαδή για κοινωνικές ενισχύσεις, για συγκεκριμένο στόλο που και επίσης αυτά τα επεισόδια με, τη, με τους πειρατές. Γιατί έχουμε στον Ειδικό ωκεανό την επιχείρηση Αταλάντη. Σας παραπέμπω στα πρακτικά του Συμβουλίου, Συμβουλίου Αλίας, γιατί εκεί συζητήθηκε το θέμα και πριν από λίγους μήνες αναλάβαμε και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ανταποκρίθηκε το Συμβούλιο Μεταφορών. Και θα συνεχίσουμε. Και γι' αυτό σας ξεκαθαρίζω. Η προσπάθεια έγινε ούτως ώστε σύντομα και υπό την αιγύδα των ε, Ηνωμένων Εθνών έχουμε κάποιο είδου προστασία στον ειδικό ωκεανό. Όπου τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί εκεί μεγάλη έκταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο τότε έγινε θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για το τι πρωτοβουλίε μπορεί να παίρνει η Ευρώπη σε ε, επίπεδο Διεθνού σκηνή για να μπορεί να βοηθήσει. Σε αυτή την περίπτωση ε, του αλληλείς, αλλά σε άλλε περιπτώσει μπορεί να βοηθήσει άλλου, άλλε δραστηριότητε. Ε, τώρα τις νέες αυτές περιοχέ. είναι συγκεκριμένο θέμα και ευχαριστώ να σας πω γιατί υπήρξε αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία είχαμε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του στόλου μας αλλά είχαμε ταυτόχρονα σε κάποιες ε, περιοχές εγκαταλείφθηκαν κάποιες συγκεκριμένες ε, αληθικές δραστηριότητες και προχώρησαν προς ένα μετασχηματισμό εκεί οι στόλοι και οι ελίες. Τώρα εντάξει είναι κάποια θέματα τα οποία άπτονται της εθνικής πολιτικής αλλά πάντως δεν έχω πρόβλημα και ό,τι, ό,τι, είχε γίνει τότε πριν πολλά χρόνια μπορώ να σας τα δώσω σαν πληροφορίες. Πάντως, οι την του στον Δικό Ωκεανό είναι αλήθεια ότι το θέμα αυτό είναι ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. για τα ευρωπαϊκά σκάφη που βρίσκονται εκεί. Και στο λέω αυτό ξεκάθαρα. Εκεί Τελείω νόμιμα ασκούνται στο του οι Ευρωπαίοι αλλιεί. Αυτό σα το λέω, να το σημειώσετε και να το ξέρετε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά οδήποτε ευρωπαϊκό σκάφος το οποίο τώρα βρίσκεται στον Ινδικό. Και το καλύτερο είναι αυτό το που μπορούμε να κάνουμε εδώ εμείς από τα θεσμικά όργανα και τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει για να συνεχιστεί η δραστηριότητά τους που είναι Ελία Πουγενή υπεύθυνο και νόμιμο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και τις εξηγήσεις που δώσατε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σταθώ ε, σε ένα θέμα που ως πρόεδρος νομίζω ότι έχω την ε, υποχρέωση να ε, σταθώ. Αναφερθήκατε στις θεσμικές σχέσεις για την εξωτερική πολιτική. Η συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί ειδικέ αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο ακριβώς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το μόνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να διασαφηνίσω είναι ότι είναι αναφέροντο δικαίωμά μας, το οποίο μας το δίνει η συνθήκη και ε, η Επιτροπή Αλίας μας εδώ σε θέματα διαπραγματεύσεων που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ούτε του Συμβουλίου λοιπόν ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εκτός λοιπόν από αυτά τα θέματα, σε όλα τα υπόλοιπα θέματα το Κοινοβούλιο ε, έχει δικαίωμα στην απόφαση. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι γίνεται στις περιφερειακές οργανώσεις αλίας και στις μικτές ε, συμφωνίες. Και επειδή συμμετέχετε ως Συμβούλιο εσείς, επομένως, πλέον το Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει το ίδιο επίπεδο συμμετοχής όπως και εσείς. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το Συμβούλιο πάντα ήταν αντίθετο σε κάτι τέτοιο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας, απλώς σας λέω για να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα και θα πάμε μέχρι τέλος προκειμένου να υλοποιηθεί. Ήθελα να το διευκρινίσω, είναι θεσμικό το θέμα, το θεωρώ σημαντικό και εσείς ως του πρώτου εξαμήνου ε, στο οποίο τίθεται σε ηχή η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να το γνωρίζετε. Θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ σαφές ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ευχαριστώ λοιπόν κυρία Υπουργή, σας εύχομαι καλή επιτυχία στη διάρκεια του εξαμήνου σας και είμαι βέβαιη ότι εσείς που προέρχεται από μια χώρα που έχει, όπως είπα και πριν, πολλά ελευτικά συμφέροντα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα της ηλεία, θα διαδραματίσετε πολύ σημαντικό ρόλο στον αλληλευτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή τύχη, καλώς ορίσατε. Αν θέλετε το λόγο, μπορείτε να παρέμβετε. Ε, μόνο το εξής, ε, κατάλαβα πάρα πολύ καλά, εσείς δεν κάνατε ερώτηση, εγώ απλώς ήθελα να χρησιμοποιήσω τα λεγόμενά σας Γνωρίζω αυτή τη συμμετοχή και για τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας και για τις μικτές επιτροπές. Αυτό προσπάθησα να διαβιβήσω και σας παρακαλώ πρέπει να είναι σαφές ότι εσείς δεν ρωτήσατε, απλώς μου το διαβιβάσατε και εγώ χρησιμοποίησα τα λεγόμενά σας μιλώντας, ε, έπιασα τα δίχτυα για να χρησιμοποιήσω και αλληλευτικούς όρους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και ε, χρησιμοποίησαμε πολύ χρήσιμο βέβαια χρόνο με την Υπουργό. Προχωράμε στο 9 τώρα που είναι η παρουσίαση μιας μελέτης για τις επιπτώσεις του ΠΟΕ και των εμπορικών διαπραγματεύσεων στον αλληλευτικό τομέα. Ε, είδατε αυτό το έγγραφο σε διάφορες μορφές και βεβαίως είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ένας από τους συντάκτες θα μας το παρουσιάσει και παρακαλώ να καθίσει, να αρχίσει την παρουσίασή του και ε, ε, όλοι να χειροκροτήσετε τον ε, συντάκτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη. Institut der Universität Wageningen erstellt haben im vergangenen ε, πρόκειται για μια μελέτη την οποία καταρτήσαμε πέρυσι. Ε, γιατί αναλύσαμε το κοινοτικό ε, δασμολογικό σύστημα εγώ βέβαια είμαι νομικός και έτσι θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το εκτενές αυτό σύστημα και την μελέτη ε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικοδομητικά σαν εργαλείο εργασίας και μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες ερωτήσεις. Η μελέτη ε, μας ανετέθη το 2008 απεφασίσει ε, το Σεπτέμβριο οπότε ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την εικόνα του Σεπτεμβρίου 2009 ε, αναφερόμαστε στον όγκο τον εμπορικό και τους εμπορικούς εταίρους και ιδίως ε, τον τομέα αλίας Ευρωπαϊκής Ενέσεως τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την αλία και μετά θα αναφερθώ σύντομα με την ε, ε, στην ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχει επιπτώσει στην αλληλεία, μετά στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και ε, τέλος τις ε, γενικές επιπτώσεις που θα είχαν αντίκτυπο εις ε, το θέμα της αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ενώσεως, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε γενικότερο και σε περιφερειακό πλαίσιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο πίνακα που παρουσιάζει ε, τις, ε, ε, τους βασικούς παγκόσμιους εισαγωγείς. Βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 17,1 δισεκατομμύρια ευρώ και οι Ηνωμένε Πολιτείε 11,2 και ε, η, Ιαπωνία και μετά έρχεται τέταρτη η Κίνα με μεγάλη διαφορά 3,3 δισεκατομμύρια. Ε, στον πίνακα αυτό βλέπετε ποιοι είναι οι βασικοί προμηθευτές η ε, ε, Νορβηγία, η Κίνα, η Ισλανδία και μετά οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Μαρόκο και βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν πολλά ψάρια τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και μετά εξάγονται ως μεταποιημένα προϊόντα. Και γι' αυτό παρουσιάζουμε εδώ παραδείγματο χάρη τον πίνακα του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Κίνα από του έτους 2000 δηλαδή κατά την τελευταία ετία, όπου βλέπουμε στη μία πλευρά τις εισαγωγές των μεταποιημένων αληφτικών προϊόντων από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξήθηκε 133% μεταξύ 2000 και 2006 ενώ συγχρόνως οι εξαγωγές από Ευρωπαϊκή Ένωση προς Κίνα για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν έξι φορές. Εξαπλασιάστηκαν δηλαδή. Ε, επιπλέον διαπιστώσαμε ότι 25% των αναγκών καλύπτονται από ε, ε, από αναπτυγμένες ε, χώρες και ότι το ποσοστό των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 30% και 60% των εισαγωγών από μη ανεπτυγμένες ε, το 60% των εισαγωγών προέρχεται από μη ανεπτυγμένες χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο βασικός εισαγωγέας αληφτικών προϊόντων ε, και αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου των ε, παγκοσμίων εισαγωγών βλέπουμε ότι οι βασικοί προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι η Κίνα και η Ισλανδία ενώ οι μη αναπτυγμένες χώρες αντιπροσωπεύουν μόνο 5% των εισαγωγών. Σχετικά με ε, τα ε, δασμολογικά θέματα βλέπετε εδώ τις ε, βασικές εισαγωγικές χώρες αλλά θα επικεντρωθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα έχουν επίσης πολύ υψηλούς δασμούς. Ε, βλέπουμε βέβαια μέσει τιμές και ε, δεν μπορούμε εδώ ε, να αποκομίσουμε ακριβείς παρατηρήσεις ε, βλέπουμε όμως ότι κατά ε, κατηγορία προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα με μεγαλύτερη αξία εισαγωγική έχουν μειότερο ποσοστό ε, και βλέπετε ότι αντιπροσωπεύουν οι, τα μη μεταποιημένα προϊόντα 9,4% και τα μεταποιημένα 9,8% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δούμε επίσης ε, πόσο κλιμακώνονται ε, οι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, η κλιμάκωση αυτή δεν είναι πολύ σημαντική και διαπιστώνουμε ότι όσο πιο μεταποιημένο είναι το προϊόν τόσο μεγαλύτερος είναι και ο δασμός για να υπάρξει ε, μια προστασία των θέσεων εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η αύξηση είναι σχετικά μικρή πράγμα το οποίο ε, ε, αντιπροσωπεύει απλώς ε, την, ε, το, τη διαφορά μεταξύ δασμών των μη μεταποιημένων και των μεταποιημένων. Ε, ε, διαπιστώνουμε όμως τον επόμενο πίνακα ότι υπάρχουν διάφορες ε, εχμές δασμολογικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες ξεπερνούν το 25% και μπορεί να είναι πολύ υψηλό το ποσοστό δασμών παραδείγματος χάνει για το πεταποιημένο τόνο σε σχέση με άλλα είδη. Βλέπουμε εδώ τις ε, ε, ε, τις προτιμησιακές μεταχειρήσεις από πλευράς δασμολογικές και ε, τα διάφορα ε, ποσοστά των ε, δασμών που επιβάλλονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τέλος πώς καταλήγουμε ε, κατόπιν εφαρμογής των προτιμήσεων βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον ότι όπου υπάρχουν κανόνες του ΠΟΕ ε, υπάρχουν και ε, περιφερειακές και τοπικές συμφωνίες αυτό το οποίο μπορείτε επίσης να δείτε στον πίνακα αυτό είναι ότι στην τελευταία γραμμή έχουμε τη συνδρομή των διαφόρων ε, εργαλείων που, προτιμησιακών που χρησιμοποιούνται στην πλήρη κατάργηση των δασμών εκ των οποίων βλέπουμε ότι η συμφωνία ε, ΕΠΑ όπως και ορισμένες διημερείς συμφωνίες ε, συνδυάζονται με μείωση των δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό ίσως οφείλεται στην ευρεία χρήση αυτού του εργαλείου διότι η, ΕΠΑΣ, η ΕΠΑ είναι διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες ε, οι οποίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Μπορούμε όμως να πούμε συνολικά ότι 25% των εισαγωγών είναι ανεφδασμών, ένα 25% έχει ε, σχετικά χαμηλούς ε, δασμούς και ε, ένα 26% επίσης ε, έχει χαμηλά, ε, χαμηλούς δασμούς κατόπιν εφαρμογής των περιφερειακών ή διμερών προτιμησιακών συμφωνιών. Εδώ διευκρινίζουμε την, την κατάσταση ανα ε, είδος ε, ψαριού και ε, αναλόγως της καταστάσεώς τους. Παραδείγματος χάρη για τον τόνο όπου έχουμε 22% Υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά με τον τόνο που συνήθως ε, ε, έχει ένα δασμό 10,9%. Θέλω να ε, συνοψίσω τώρα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικά υψηλούς δασμούς και ορισμένες μάλιστα εχμές ε, για τα, τον τόνο και ε, για τον αστακό και διαπιστώνουμε ότι το η αύξηση ε, στο σύστημα αυτό δεν είναι πολύ σημαντική ε, αλλά θα ήθελα εδώ ε, να σας πω ότι υπάρχει μία απαρίθμηση των άλλων των μη δασμολογικών εμποδίων το οποίο δεν πρέπει να αναλυφθεί ως κριτική απλούστατα αναφέρω τις διάφορες ρυθμίσεις οι οποίες επηρεάζουν τον τομέα της αλληλείας βεβαίως ε, το, ουσιαστικά ο πρώτος λόγος υπάρξεων των ρυθμίσεων αυτό είναι η διατροφική ασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων, επίσης οι ανάγκες σημάνσεων όπου ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα που συνοδεύουν ε, τα, τα λιεύματα και ε, επιπλέον βλέπουμε άλλες ρυθμίσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως που επηρεάζουν το αληφτικό εμπόριο και ουσιαστικά την σχέση της ε, ε, μειώσεως των δασμών με ε, την ύπαρξη των μη δασμολογικών εμποδίων διότι βλέπουμε ότι από το έτος 2000 μέσω των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΗ τα ρυθμιστικά, οι ρυθμιστικοί κανονικοί έχουν διπλασιαστεί Ε, υπάρχει ε, διαφορετική εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε διάφορα κράτη πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια πιο χαλαρή εφαρμογή των κανονισμών και ε, δημιουργεί μια στρέβλωση η οποία επηρεάζει το εμπόδιο. Τώρα ερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ όπου υπάρχουν τρεις θεματικές ενότητες που είναι σημαντικές για την αλληλεία. Καταρχήν το θέμα της μειώσεως των δασμών χάρη στο ΝΑΜΑ, δηλαδή εις τις διαπραγματεύσεις προσβάσεως στις μη γεωργικές αγορές επίσης εις ε, τις ε, επιδοτήσεις της αλληλείας και εις ε, εργαλεία για την προστασία του εμπορίου. Βεβαίως είναι προφανές ότι δεν ε, υπάρχει η ισότιμη αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αλληλευτικών προϊόντων και βιομηχανικών προϊόντων το τομέας των οποίων έχει τελείως διαφορετικά συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι όλα τα προϊόντα τα οποία λαμβάνονται υπόψη στα ΝΑΜΑ ε, ε, αποβλέπουν σε μία μείωση των δασμών και στην κατάρτιση ενός κοινού δασμολογικού επίπεδου και στην αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προσπαθήσει να εξαιρέσει τα αλλιευτικά προϊόντα από αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, ε, δεν ακολούθησε αυτή τη γραμμή εις ε, τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και τον τελευταίο καιρό έχουν εφαρμοστεί υψηλοί συντελεστές που βασίζονται στον ελβετικό υπολογισμό, ο Swiss Formula, όπου υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές για ανεπτυγμένες και υποανάπτυξη χώρες 8 και 20, 22 ή 25. Και αυτό ε, δίνει διάφορες δυνατότητες να εφαρμοστούν επίσης και εξαιρέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ε, το ποσοστό του 8% πρέπει να αποτελέσει στόχο αντί για το ισχύον 15% ε, για μία σειρά προϊόντων τα οποία είναι ευαίσθητα. Βλέπετε όμως ότι ε, δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή και λόγω πιέσεως χρόνου δεν ε, ε, προχωράνε τα θέματα. Ένα άλλο θέμα που, στο οποίο εστιάζονται οι διαπραγματεύσεις είναι ε, ε, η κατάρριξη προτιμήσεων και υπάρχει ε, μη μία πρόταση να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τα, τους υψηλούς δασμούς για την επόμενη πενταετία στον τομέα μάλιστα της αλίας αυτή η επέκταση λαμβάνοντας ε, η υπόψη ε, το γεγονός ότι οι προτιμήσεις είναι ένα μέτρο για να μπορέσει κανείς να προσαρμοστεί στις αλλαγές ε, δείχνει ότι σε ορισμένες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ε, διεκόπησαν αναφερόντουσαν ε, εις ε, τους τομείς που συζητούνται με τις Ηνωμένε Πολιτείες και δεν ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να υπάρξουν τομεακές διαπραγματεύσεις για μείωση ε, των δασμών ε, διότι δεν, δεν προχωράει το θέμα αυτό. Τέλος, ε, έχω να προσθέσω ότι βάσει αυτών των στοιχείων ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές διευκρινήσεις οι οποίες επιπλέον χρειάζονται διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επεμβαίνει σε ευαίσθητους τομές όπως η Σαρδέλα και ο τόνος και ε, εφαρμόζει τα βατικά μέτρα τα οποία μπορούν να καλύψουν μία δεκαετία. Επίσης θα πρέπει να λεχθεί ότι δέχεται το ποσοστό των χωρών εκτός χωρών και να χαθεί υπέρ ε, των ασιατικών συμφερόντων προς όφελος των ασιατικών συμφερόνων. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, ε, ε, υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις για να αποφύγει κανείς τις αρνητικές επιπτώσεις της αλίας, δηλαδή υπεραλίευση ε, και υπάρχει συγχρόνως μία απαγόρευση για ε, την... Ε, υπάρχουν επίσης μέτρα τα οποία αναφέρονται ε, σε, σε έναν εξυγχρονισμό του στόλου σε διάφορες βαθμίδες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λαμβάνει μέτρα τα οποία προσπαθεί να μειώσουν ε, τον υπερβολικό αριθμό αλλευτικών σκαφών ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι οι επιδοτήσεις στα πλαίσια των ε, αλλιευτικών ε, συμφωνιών που ε, δίδονται εις τον κοινοτικό στόλο αλλά δεν ξέρουμε εάν θα μπορέσει αυτό το σύστημα να συνεχίσει να ισχύει εάν αναθεωρηθούν οι συμφωνίες άλλα μέτρα είναι οι προστατευτικές ρήτρες και τα ε, μέτρα anti-dumping που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια ε, του γύρου της Ντόχα βλέπουμε ποιες είναι οι διαδικ... ποια είναι τα δικαστικά στοιχεία, ε, ε, γίνονται έρευνες για απόδειξη ότι ε, υπάρχει dumping για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα μέτρα καταπολέμησης του dumping αλλά υπάρχει μία σαφής τάση ότι επιζητείται μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, μία μεγαλύτερη εμπλοκή των ε, ενδιαφερομένων βιομηχανιών κατά τρόπον ώστε ε, να ε, εφαρμοστεί σωστά η συμφωνία και να, ε, και να συνδυάζεται και με τα συμπεφωνημένα στον ΠΟΕ. Τέλος, όσον αφορά τις περιφερειακές και διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώσαμε ε, μιλώντας για την ε, μείωση των δασμολογικών ποσοστών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει περιφερειακής και διμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες με πέραν των 120 χωρών και και ε, ότι ε, υπάρχουν συγχρόνως και προτιμησιακές συμφωνίες με διάφορα ε, κράτη-μέλη του ΠΟΕ η δε τάση αυτή θα συνεχιστεί εφόσον δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις του γύρου της ΔΟΧΑ. Εν μεταξύ Υπάρχουν ε, διάφορες θεματολογικές ενότητες οι οποίες αναφέρονται ή στις ε, προτιμήσεις ε, τις οποίες χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως μία συμφωνία ελευθέρου εμποδίου με τη Νότιο Κορέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή ε, του, της συνθήκης αυτής να μειώσει και να καταργήσει ε, τους δασμούς ε, πράγμα το οποίο βρίσκει αντίθετο τον ενδιαφερόμενο κλάδο ή στην Ευρώπη υπάρχουν διαπραγματεύσεις ε, για συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις ε, χώρες του Μερκοσούρ που δεν προχωράνε ε, διαπραγματεύσεις με την Κεντρική Αμερική που έχουν διακοπεί και με την κοινότητα Αντέαν συνοψίζοντας τελικά θέλω να ε, εξετάσω τα αποτελέσματα από το πρίσμα της δασμολογικής δομής διαπιστώνουμε ότι από την Ασία ιδίω για την υδατοκαλλιέργεια αντιμετωπίζουμε προβλήματα γιατί υπάρχουν ε, ε, ανεπτυγμένες μεταπητικές βιομηχανίες την Κίνα και ε, την Ασία γενικότερα και ε, ε, αν υπάρξει κατάργηση των δασμών οι τιμές εισαγωγής των προϊόντων αυτών θα μειωθούν περαιτέρω και μακροπρόθεσμα ε, θα δημιουργηθεί μία κατάσταση ε, όπου η χώρες ε, ΑΚΕ που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στις κοινοτικές αγορές θα χάσουν ένα σημαντικό μέρος ε, της αγοράς που καταλαμβάνουν. Ε, θα υπάρξουν όμως τομείς όπου θα συνεχίσουν να υπάρχουν υψηλοί δασμοί και θα μπορέσουν να επηρεάσουν επίσης την ε, ε, γενική κατάσταση. Όσον αφορά την ε, μείωση των προτιμησιακών ρυθμίσεων για παραγωγούς από τις λιγότερα ανεπτυγμένες χώρες αυτές θα είναι εις βάρος των χωρών και ελπίζω ότι τα στοιχεία που σας παρουσίασα σας ήταν χρήσιμα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Ε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μου δώσατε. Στη συνέχεια, έχει ζητήσει το λόγο. Ποιος? Η κυρία Λέβιν. Μα έτσι δεν που το χέρι. Καλά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το τόσο μας είπατε. Ευξανόμενες εξαγωγές δηλαδή, από την κοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως και μας αναλύσατε το τι γίνεται με αυτή την ε, επανεξαγωγή που γίνεται. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για ελεύθερα είδη. Μήπως ε, μιλάτε για προϊόντα υδατοκαλλιεργία. Πρέπει να σας πω ότι η μελέτη αυτή έχει γίνει από ένα Ινστιτούτο και μπορώ να βασιστώ στα στοιχεία. Ε, η μελέτη όμως αυτή αναφέρεται σε στατιστικές ε, δεν ξέρω τι ε, ροές κρύβονται πίσω από τα στατιστικά στοιχεία εάν πρόκειται δηλαδή για εισαγωγές, μεταποιήσεις και ε, μετεξαγωγές των ε, προϊόντων που εισήχθησαν αρχικά σε ακατέργαστη μορφή. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εισήγησή σας. Ε, κοιτάω τώρα, ρίχνω μια ματιά και τα συμπεράσματα. Για πέστε μας. Στα πλαίσια της ελευθερικής αστριότητας, ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι Ευρωπαίοι. Τι γίνεται όσον αφορά τους δασμούς και τις συνέπειες της απορρίθμισης. Ποιοι είναι οι κλάδοι, οι τομείς, ε, τα κομμάτια της δραστηριότητα που είναι οι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Άκερ ιδιαιτέρως ο, ο τόνος η σαρδέλα και η γαρίδα. Και εγώ λέει πρώτος, θέλω κάτι να σας πω. Ο τόνος. Όπως ξέρετε, είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, η αλλαγή των δασμών, η τιμολογική πολιτική στη διεθνή αγορά. Μας μιλήσατε λίγο γι' αυτά, αλλά για πέστε μας. Έχετε λάβει υπόψη σε συγκεκριμένο τρόπο το ότι όσον, όσοι επιτοπλίστων μεταπημένος τόνος περισσότερες αγωγές μας τέλος πάντων έχουν κάποια, κάποιο προτιμησιακό καθεστώς για τους δασμούς. Είναι χώρες ακέ, όπως ε, και εσείς είπατε. Ταϊλάνδη, άλλες χώρες της ε, Ανατολής από όπου εισάγουμε. Οπότε αυτό θίγει όχι μόνο τις χώρες ΑΚΕ αλλά και τους κοινωτικούς ε, αλίες. Επομένω, ε, δεν πρόκειται εδώ για τον δασμό το οποίο είπατε. Είναι πολύ φτηνότεροι οι δασμοί. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΟΕ, αυτές τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις και την κατάργησή τους. Και από στιγμή που θα έχουμε μια μεταρρύθμιση που να γίνει όπως πρέπει, δεν θα χρειάζονται επιδοτήσει Να είναι δηλαδή ένας κλάδο αυτοχρηματοδοτούμενο. Επικερδή. με σωστούς κανόνε παιχνιδιού. Οπότε δεν έχω πρόβλημα με αυτή την κατάργηση. Όμως υπάρχει ένα αντάλλαγμα που είναι οι επενδύσεις σε τρίτες χώρες, ε, όπου έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς περιορισμούς που δεν ξέρει, δεν γνωρίζει άλλη αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα. Ε, πώς μας ήταν να κόψουμε τις επιδοτήσεις και αυτοί από την άλλη μεριά ε, έχουν τις, ε, τους περιορισμούς. Άρα, να μειώσουμε με τις επιδοτήσεις και αυτοί να μειώσουν τους περιορισμούς. Να κάτσουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο θέματα. περικοπή των επιδοτήσεων και ταυτόχρονα άνοιγμα των ε, αγορών για επιδοτήσεις στις τρίτες χώρες. Χιλή όπου, όπου στο καλό είναι. Εγώ δεν ήθελα τίποτα να σας πω, ίσως κάποιος άλλος να λάβει το λόγο για να λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως αν μπορείτε, πέστε μας. Έχετε το λόγο. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, Θεωρητικά βέβαια διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, εφαρμοσμένων ε, και ονομαστικών ε, ποσοστών δασμών και ε, ε, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι πολύ αισθητή. Ουσιαστικά όμως ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες όπου ισχύουν ακόμη τα υψηλά ποσοστά δασμού αλλά δεν μπορώ να σας εξηγήσω σε ποιες χώρες ισχύουν αυτά τα συστήματα όσον αφορά ε, τις ε, μειώσεις ε, των δασμών εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη χρήση χρηματικών στηματικής στήριξης ε, μέσα στα πλαίσια της preferential ε, tariff treatment που ισχύουν για τις υποανάπτυξη χώρες ε, υποθέτω ότι μπορεί να δημιουργήσουν όντως διαφορετικά. Θα ήθελε κάποιο άλλο βουλευτή το λόγο. Ήθελα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μιλάτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τον κύριο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο που προέβη στην εισήγηση. Και θα θέλαμε απλώς να σας πούμε ότι συναρμόδιας είναι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Αλίας που τους εκπρόσωπω. Οπότε και όταν χρειαστεί θα δώσω τη σκητάλη στο συνάδελφο που ασχολείται με τα εμπορικά. Απλώς. Θα σα πω ότι είναι κρίμα που ποτέ δεν μας συμβουλεύτηκαν οι σύμβουλοι. Α πούμε αυτό το οποίο κυρία Λέβιν όσον αφορά την ε, επανεξαγωγή των προϊόντων Ελίας που υφίσταται αυτή την ε, ε, μεταποίηση στην, στην Κίνα και έχουμε και την επιβάρυνση όσον αφορά το γιατί έχουμε τα ψάρια τα οποία τα ψαρεύουν. Οι Νορβηγοί πάνε στην Κίνα και κατόπιν επανεξάγονται στις ευρωπαϊκές αγορές. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη και είναι ζωντανή, είναι, σαν, μελέτη που έγινε επιτόπου, μας δίνει αυτά τα στοιχεία για το τι γίνεται σε διάφορα σημεία και στην Ισλανδία έχουμε αυτές τις μεγάλες εξαγωγές αγορές τις πιο μεγάλες του κόσμου όπως αναφέρθηκε στην ε, έκθεση οπότε και έτσι αναλαμβάνουμε και εμείς μια μεγάλη ευθύνη όσον αφορά την ε, παγκοσμία διακυβέρνηση και διαχείριση της αλίας θα πρέπει η αγορά μας να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ασκήσουμε κάποια επιρροή στην παγκόσμια διαχείριση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη αλληλεία. Και γι' αυτό το λόγο και σας λέω ότι είναι κρίμα ότι έχουμε αυτή την παρουσίαση του Αγίου, του κανονισμού και του κανονισμού που αφορά την υγεία των καταναλωτών που αναφέρθηκαν εδώ ως φραγμή προς το εμπόριο. Μη δασμολογική φραγμή του εμπορίου. Η πρόταση στασία της υγείας δεν αποτελεί μη δασμολογικό φραγμό στο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και για τον ε, κανονισμό Αγίου. Η θέση εμπορία στην κοινωτική αγορά κάποιων ε, προϊόντων λαθρελίας. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το διεθνές εμπόριο. Όπως και οι κανόνες της προέλευσης που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι ούτως ώστε να ισχύσει η θεσμολογική πολιτική. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε όλα αυτά να τα θεωρήσουμε ως μη δασμολογικούς φραγμούς πρόκειται για κάποιους φραγμούς που συχνά δημιουργούν οι εταίροι μας. Η απαγόρευση ας πούμε εξαγωγών από τον Καναδά επίσης ε, ε, κάποιες ε, επιβαρύνσεις της Ισλανδίας εις βάρος αλληλευτικών ευρωπαϊκών. Επίσης, προτεθώ και να πω δύο λόγια για την επιδότηση σε σχέση με τη μεταρρύθμιση κιόλα, που είναι κάτι που μας απασχολεί, διότι στα πλαίσια της μεταρρύθμισης ακόμα δεν τα έχουμε βρει μεταξύ μας όσον αφορά την πολιτική των επιδοτήσεων που θα ακολουθήσουμε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ελίας. Γιατί έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν οι επιδοτήσει όσον αφορά τη δραστηριότητα αυτή. Και Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ελία που είναι κλάδο ποιος ακόμα δεν έχει σταθεί στα πόδια του, είναι αρκετά εύρωστο ούτω ώστε να μπορέσει να αντέξει μια πλήρη και άμεση αποκέντρωση και απελευθέρωση όπως προτείνεται. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του ΠΟΕ να έχουμε μέτρα για τις επιδοτήσεις, τα οποία όμως να βασίζονται σε κοινοτική συνένεση. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει ταχαίως. Επίσης ελπίζουμε ότι τα μέτρα τα οποία θα λάβει ο ΠΟΕ να μην απελάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως σήμερα προτείνεται. Έτσι θα, έχουμε την Κίνα ως πρώτη εξαγωγική δύναμη. Μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στην Αλία η οποία θα μπορεί να επεκταθεί από πλευρά παραγωγή χωρί να έχει καμία επιβάρυνση. Αυτό δεν μας συμφέρει. Ούτε έχει καμία σχέση με την προστασία της Ελίας παγκοσμίω. Απλώς έχω να σας πω ότι από πλευράς μας θεωρούμε ότι το, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί η κοινωνική πολιτική καλύπτει τα μισά από τα ψάρια που καταλώνουμε, ενώ η εμπορική πολιτική τα καλύπτει όλα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και επίση ε, ευχαριστώ με οποιοδήποτε συνάδελφο της Επιτροπή να συνοηθούμε για να βοηθήσουμε, να διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και για την εκθεσή σας. Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να είχαμε συζητήσει το θέμα της οικολογικής επισήμανσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αγιογωγές και η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει στις ε, παρουσιάσεις από πλευράς ε, προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το εμπόριο θα μπορούσε να είναι μια καλή άγουσα για την βιωσιμότητα των πόρων είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που είναι αυτή τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την υπόθεσή σας. Ε, ολοκληρώσαμε το σημείο 9 τώρα. Περνάμε στο σημείο 10, το καθεστώς των εισαγωγών των εισαγωγικών προϊόντων και των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας η είναι ο κύριος Καντέκ, θα του δώσω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ε, στη συνέχεια με την προηγούμενη παρουσίαση θα συζητήσουμε για πρώτη φορά αυτή την έκθεση. Η πολιτική μου ομάδα και εγώ σας προτείνουμε αυτή την ε, ε, κατά πρωτοβουλία έκθεση λόγω της σημαντικής σημασίας του θέματος το οποίο πραγματεύεται και βλέπουμε ότι καταρχήν συνδέεται με το, την έκθεση για την πράσινη βίβλο και την ε, έκθεση για τη στρατηγική για την ε, ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια γι' αυτό και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ασχοληθούμε ε, και πιο συγκεκριμένα με αυτό το θέμα διότι όταν εξετάζουμε το καθεστώς των εισαγωγών αλληλευτικών προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ένας ανταγωνισμός με τα προϊόντα της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν εξετάζει κανείς τον τομέα της ε, ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είδαμε τι μπορεί να συμβεί με την Κίνα παραδείγματος χάρη. Οι αριθμοί είναι εύγλωτοι ότι ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο σημαντική αγορά εισαγωγική για τα προϊόντα της αλίας και, την υδατο... και τις ε, πριν και από τις Ηνωμένε Πολιτείες εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τις εισαγωγές ώστε η ε, παραγωγή κοινοτική αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει λιγότερο από 23% δηλαδή ε, έχουμε 77% εισαγωγές το οποίο είπε και η κυρία Δαμανάκη την περασμένη εβδομάδα μίλησε για 70% και ουσιαστικά έχουμε 77% των εισαγωγών προβλέπετε ότι θα υπάρξει μέχρι το 2030 ακόμη αύξηση κατά 1,5 εκατομμύριο και όλες ε, αυτές θα είναι εισαγωγές ε, οι οποίες παρόλα αυτά δεν θα καλύψουν την ε, ζήτηση και οι εισαγωγές καλύπτουν διαφοροποιημένες και περίπλοκες ανάγκες. Ανησυχούν όμως τους ενδιαφερόμενους από τον κλάδο και γι' αυτό θέλω στην έκθεσή μου να παρουσιάσω αυτές τις ανησυχίες ε, βασίζομαι ουσιαστικά σε τρεις πολιτικές σκέψεις και θα σας τις παρουσιάσω καταρχήν και μετά θα τις συγκρίνω με την πραγματικότητα. Ε, η πρώτη μου ιδέα είναι ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται ε, έχουν παραχθεί υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ισχύουν εις ε, την κοινότητα και υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δείξουμε πώς αυτό επηρεάζει τους Ευρωπαίους παραγωγούς Επίσης, δεδομένου του κοινού εξωτερικού δασμολογίου που είναι πολύ χαμηλό αλλά μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες τομείς, παραδείγματος χάρη τον τόνο ή τη σαρδέλα, ε, υφίσταται ορισμένες πιέσεις καταρχήν όσον αφορά τις μη αγροτικές αγορές ε, στον ΠΟΕ και ε, ετοιμάζονται να μειώσουν την προστασία αυτή ενώ τα γεωργικά προϊόντα είναι της αποτελεσματικής αρμοδιότητος του Επιτρόπου Γεωργίας τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν καλύπτονται καθόλου. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την έκθεση κατά πρωτοβουλία θέλω να τονίσω ότι η πράσινη βίβλος δεν αναφέρεται ή στις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Απλούστατα σε μία παράγραφο στη σελίδα 19 υπάρχει μία απλή μνήα χωρίς να λέει ότι οι ε, μειώσεις που θα επιβληθούν εις τους, ε, ε, εις, εις τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα οδηγήσει σε μία σημαντική μείωση και ότι το ποσοστό το οποίο θα μειωθεί θα καλυφθεί από εισαγωγές από εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί λοιπόν να υπάρξουν θυσίες για τους δικούς μας παραγωγούς ε, αν πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές από προϊόντα που δεν παράγονται από τις ίδιες συνθήκες. Δεν θα ήταν καλύτερα η ε, ευρωπαϊκή αγορά να, η, να μην υποκινεί τις τρίτες χώρες να υπεραλλιεύουν διότι εμείς αντιπροσωπεύουμε απλούστατα 6% της ε, συνολικής ε, ε, αλευτικής δυνατότητος γιατί λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει όλες τις ευθύνες. Αφού λοιπόν εξετάσαμε τα συμφέροντα των μεν και των δε θα ήθελα να διατυπώσω συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική, αγορά, ε, μελλοντική οργάνωση της αγοράς της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας ε, διότι οι ε, παρακλήσεις μας δεν έχουν ίσα ακουστεί και ε, πολύ φοβούμαστε ότι οι διαπραγματευτές θα απεμπολίσουν τα συμφέροντά μας και γι' αυτό θα ήθελα να έχω τις γραπτές και προφορικές σας προτάσεις. Θα σας ενημερώνω σε όλα τα στάδια της κατάρτισης του σχεδίου εκθέσεώς μου για την πρόοδό μου. Ξέρω το θέμα αυτό ενδιαφέρει πολλούς από εσά, ιδίω μέσω πολλών ερωτήσεων που ετέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην υποψήφια επίτροπο κυρία Δαμανάκη σχετικά με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και παρόλο που γενικώ τα πήγε πολύ καλά δεν νομίζω ότι απάντησε καλά τουλάχιστον κατά τη δικιά μου κρίση. Ε, οι εργασίες λοιπόν που θα διεξάγω θα βασιστούν στις μελέτες του ΠΟΕ που έχουν καταρτιστεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσης. Επίσης ε, απευθύνω συγκεκριμένα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διάφορες ε, αγοράς, υγείας, θα κάνω συναντήσεις με τους, με τους εκπροσώπους των διαφόρων υπηρεσιών, θα υπάρξει διαβούλευση με τους αλληλείς και τους υπευθύνους υδατοκαλλιέργειες και ε, διανομής και εμπορίας διότι θα πρέπει να καλύψουμε όλες ε, τις ε, απόψεις στη συνέχεια στις Βρυξέλλες και στη Γενέβη θα ήθελα να συζητήσω με τους βασικούς εκπροσώπους των χωρών που εισάγουν προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και ε, συγχρόνως ε, συνεχώς θα είμαι με επαφή μαζί σας για να γνωρίζω ποιες είναι οι εθνικές ευαισθησίες ε, και οι προσωπικές σας απόψεις στις διάφορες χώρες σας. Ελπίζω να έχω ολοκληρώσει την έκθεσή μου μέχρι το καλοκαίρι. Σήμερα ήταν η πρώτη, είναι η πρώτη ανταλλαγή. 15-16 Μαρτίου θα έχουμε δεύτερη ανταλλαγή απόψεων κάποιο έγγραφο 7-8 Απριλίου ακρόαση για την αναμόρφωση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής 3-4 Μαΐου παρουσίαση της εκθέσεως και καθορισμός της προθεσμίας των τροπολογιών επιτροπή, ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Ιούνιο και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με την έκθεση αυτή και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να διατυπώσετε παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καδέκ. Καταρχάς, να κάνω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ε, προκύπτει και από την παρέμβαση της κυρίας Σπινόσα σήμερα το πρωί. Ε, η κυρία Σπινόσα είπε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής ε, τα προγράμματα ε, επικαιροποίησης της αρχικής, της υφιστάμενης ε, νομοθεσίας έχουν ολοκληρωθεί και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις νέες προτάσεις και τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι απόψεις σας και οι προτάσεις σας, διότι αυτό μας είπε η Υπουργό σήμερα το πρωί και νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον ο κύριος Καντέκ να γνωρίζει ποια ε, είναι αυτά τα οποία φρονείται για την μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση και θα ήθελα να κάνω και εγώ μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη Δευτέρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος συζήτησε το θέμα αυτό για την γνωμοδότησή τους ε, για την οχθεοκαλλιέργεια. Αυτή τη στιγμή εισάγονται 65.000 ε, τόνοι ψαριού παγκράσιους. Mm τα σούπερ μάρκετ μας στις 27 χώρες μέλη με διάφορα ονόματα, ε, βιετναμέζικος γάδος, ε, πάγκα, και διάφορα άλλα ονόματα. Πρόκειται για ένα ε, ψάρι χωρίς ε, κόκαλο, ε, άνοστο σχετικά, αλλά αν προσθέσουμε διάφορες σάλτσες γίνεται πολύ δημοφιλές και τιμάται και σε τιμές που... υποσκάπτουν ακόμα και τα φρέσκα αλλιεύματα που έχουμε στις θάλασσες. Άκουσα πολλούς αλληλείς να διαμαρτύρονται ότι πέφτουν οι τιμές των δικών τους ψαριών, ε, των αλλιευμάτων τους, ε, λόγω του ανταγωνισμού από το Παγκάσιους. Είμαι υπέρ του θεμητού ανταγωνισμού, αλλά αυτό το ε, προϊόν παράγεται στο δέλτα του Μήκον που είναι ένας από τους πιο μολυσμένους ποταμούς που υπάρχουν. Από ένα δείγμα που ελήφθη στην Ισπανία διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν ε, ακόμα και αρσενικό σε κάποια περίπτωση. Επίσης διάβασα και σε κάποια ιστοσελίδα ότι η τεράστια λευτική παραγωγή που έχουμε στο Βιετνάμ στις ηχθειοκαλλιέργειες ε, χρησιμοποιούνται και ορμόνες ε, οι οποίες ε, λαμβάνονται από έγκυες γυναίκες και μάλιστα από τα ούρα εγγύων γυναικών λέει ο μιλητής και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούνται σε ενέσιμη μορφή και ε, γίνεται ένεση στα ψάρια για να αυξηθεί ο αριθμός των ε, αυγών και να αυξηθεί και η ταχύτητα ανάπτυξης ε, του ψαριού αυτού. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο συχνά έχουν πάει στο Δέλτα του Μήκον για να ε, επιθεωρήσουν την παραγωγή εκεί, τι δείγματα έχετε πάρει από αυτό το ποταμό, πόσο συχνά πηγαίνετε, πότε σκοπεύετε να κάνετε την επόμενη επιθεώρηση και κατά πόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το ψάρι είναι ασφαλές και μπορούν να το καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι. Ε, διότι αυτό είναι ο αθέμητο ανταγωνισμός που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο κ. Καντέκ στην έκθεσή του. Και πρέπει να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν μα είχε πει ότι το βόλιο κρέα από τη Βραζιλία ήταν ασφαλέ και τελικά έγινε μια ανεξάρτητη έρευνα από γεωργού, από κτηνοτρόφου από την Ιρλανδία που πήγαν στη Βραζιλία, επισκέφτηκαν κτηνοτροφικέ μονάδε και διαποστάθηκαν ότι καθόλου ασφαλέ δεν ήταν και τελικά είχαμε απαγόρευση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ίδια θα γίνουν και τώρα. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τι έχετε να μα πείτε επί του θέματο. Ευχαριστώ, κυρία Λεβίν. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάντεκ για την εισήγησή σας. Με μεγάλη μου χαρά είδα αυτό τον ε, πίνακα που λέει ποιες είναι ποιες είναι οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις ε, εισαγωγές. Κίνα, Ισλανδία, ΙΠΑ, αυτή είναι η βασική εισαγωγή. Και βέβαια είπα με την Κίνα πρωταγωνιστούν, το ξέρουμε, γιατί και όλοι αυτοί και η Ισλανδία επιβάλλουν ε, πάρα πολύ σκληρούς κανόνες και αντίστοιχα σε σχέση με τις δικές μας ίδιες εργασίες είναι πολύ αυστηρή. Έχουμε εδώ πέρα ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει προσεκτικά να το εξετάσουμε και επίσης πρέπει να σας τονίσω ότι η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Κίνα είναι χώρες που έχουν ε, καταφέρει να αντιστρέψουν την φθήνουσα τάση των ε, αλιευτικών πόρων. Επομένως, εκεί οι ληφτικοί πόροι θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το 1995 και μετά αντίστρεψαν αυτή την τάση στη ΣΥΠΑ που, που, που οι πόροι ε, έδειχναν να φθήνουν με απελπιστικούς ρυθμούς. Δεν ξέρω αν είσαι μαζί μου κύριε Καντέκ. Ε, από ό,τι ξέρω συμφωνείτε. Και επίση θα συμφωνείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να τα πάμε καλύτερα στον αφορά πόρους στην Ευρώπη. Να δούμε τι γίνεται, τι αλλιεύματα με τη δεκαετία του 70, τι έγινε εδώ, στο Κάτιγκατ, όπου είχαμε 25.000 τόνους τη δεκαετία του 70 και τώρα έχουν πολύ λιγότερα. Και μιλάω μόνο για τη Σουηδία, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Βαλτική. Επομένως βρισκόμαστε σε κρίση και αυτό αφορά τους πόρους μας, γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να εστιαστούμε στο πρόβλημα γιατί βεβαίω και προβαίνουμε σε εισαγωγέ. όμως θα πρέπει κάτι να γίνει και με την οικολογική ετικέτα, το σήμα, θα πρέπει να έχουμε ανιχνευσιμότητα. Τι γίνεται με αυτά τα ψάρια από την Κίνα, θα πρέπει να ξέρουμε από πού και που έρχονται. Το ίδιο αφορά και το ποτήμα του άνθρακα. Πάει ο Σολομός στην Κίνα, ξαναγυρίζει. Ε, φυσικά και αυτό δεν είναι καλό για το περιβάλλον όμως. Ξέρω ότι έχουν γίνει αναλύσεις όσον αφορά το αποτύπωμα και στα Ιναλία. Όμως θα πρέπει να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Στη θάλασσα, ε, στη διαδρομή του ψαριού μέχρι το πιάτο. Ξέρουμε ότι ακριβώς τα ληφτικά σκάφη ε, δημιουργούν φοβερό αποτύπωμα ανθρακά. Η πρώτα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να είσαστε σε ερωτήσεις λίγο σύντομη γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να προλάβουμε την ημέρηση διάταξη σήμερα. Καπούλα Σάντος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα απλώ να πω στον κύριο Καντέκ, μια που είμαι και σκιώδη ηγητή για του σοσιαλιστέ, είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ μαζί του. Συμφωνώ με τις τρεις του προτάσεις όσον αφορά την ε, μεθοδολογία που προτείνει. Επίσης νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη μελέτη αυτή, την έκθεση αυτή, με κάποια ανάλυση, με κάποια, με κάποια, έκθεση των αιτιών της συρρήκνωσης των πόρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί όλα τα άλλα προβλήματα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θέλουμε τώρα να ξεκινήσουμε. Είναι κάτι το οποίο ε, αφορά όλα τα θέματα της έκθεσης. Οπότε, κύριε Καντέκ, εδώ είμαι. Όποτε θέλετε, στο πλάι σας να συνεργαστούμε, να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλάν Σαντέκ για την έκθεσή του γιατί ε, φέρνει ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ στην Ευρώπη και σαν καταναλωτές. Όταν ε, αναπτύσσεται μία αγορά υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση. Δεν μπορούμε εμείς να προμηθευτούμε αυτά που θέλουμε διότι το μια μας λένε είναι χειμώνας, αυξάνει η τιμή του ψαριού μετά λένε α, θέματα υγείας αυξάνει η κατανάλωση του ψαριού υπάρχουν πολλά θέματα και ίσως κάποιος θα έρθει και θα πει για να προστατεύσετε το, το, δάσος θα πρέπει να τρώτε περισσότερους σκίους. Αυτό το λέω για σκίο για Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορούμε να οργανωθούμε για να έχουμε σωστή προμήθεια για τις ανάγκες μας και ε, επίσης για το εσωτερικό ΑΕΠ της Ευρώπης δεν πρέπει ε, να αναφερόμαστε ε, μόνο εις την πρώτη ύλη αλλά και στη μεταποίηση όπου οι επιδόσεις μας βελτιώνονται όσον αφορά την αγορά. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η κατανάλωση. Πού είναι οι πόροι μας και ποιοι είναι οι πόροι μας. Επίσης ε, την, ε, και τον κεκαλυμμένο ανταγωνισμό που αναφέρει ο συνάδελφος και που είπε και ο, ο παρουσιαστής της μελέτης πού είναι η προστασία του καταναλωτού όταν εισάγουμε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας από την Ασία όπου και εκεί υπάρχει αθέμπτος ανταγωνισμός. Ευχαριστώ κυρία Γκρόμπερτ, ο κύριος Ευχαριστώ. Και εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεση διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική ίσως πρόκειται για μία έκθεση κλειδί για το μέλλον της αλίας και ε, για την ε, οικονομική κατάσταση του τομέα ε, πρέπει να εξετάσουμε την ανάπτυξη της αλληλείας στην Ευρώπη και ε, τι παράδειγμα θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη κατά τρόπον ώστε ε, το, βλέπουμε ότι ο βακαλάος όταν αγοράζεται από τον Αλιέα κοστίζει ένα, κιλό το, ένα ευρώ το κιλό ενώ στο, στο έμπορο ψαριών πληρώνεται ε, πέντε ευρώ. Αν το προσαρμόσουμε σε ψάρια τα οποία εισάγονται από τον Μεκόγκ ή από την Κίνα πληρώνουμε 2 ε, ή 5 ευρώ. Ποιος ξέρει τι πληρώνουν ε, οι, αυτοί που τα εισάγουν. Μιλάμε για θέμα το ανταγωνισμό. Ζητήσαμε από έναν από τους ε, συνεργάτες μας τι μπορούμε να κάνουμε με την κατάσταση που υπάρχει και μας απέντησε φαταλιστικά να προσαρμοστείτε. Κύριε Καντέκ, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν σκοπεύω να προσαρμοστώ. Θα πρέπει ε, η αρχική τιμή να είναι ε, αποδοτική ήδη για τον ψαρά και αν είναι αποδοτική για τον ψαρά θα μπορέσει να έχει ένα κέρδος και ο μεταποιητής και όλοι οι κρίκοι της αλυσίδος θα έχουν καλή απόδοση. Ε, επίσης ακούσαμε πριν από λίγα από τον επισκέπτη μας που μιλούσε για τον ΠΟΕ και για το διεθνές εμπόριο ότι υποθέτουμε ότι στην Ισπανία καθυστερεί η διαδικασία αντιντάμπικ και ε, ελπίζουν ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι πιο χρήσιμο αλλά εγώ θα στηρίξω την έκθεση του κυρίου Καντέκ. Ξέρει, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αλλιώς ο κύριος Μιλά για να απαντήσει. Merci, Madame la Présidente. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχίζω για το Παγκάσιο. Βλέπω ότι όσον αφορά τα υγειονομικά, μερικοί συνάδελφοι από εδώ δεν μα εμπιστευτούν τόσο πολύ. Να σα απαντήσω με συγκεκριμένα στοιχεία και σα ε, διαβεβαιώ ότι στο Βιετνάμ πάνε τακτικά οι αρμόδιοι συνάδελφοι. Πρόκειται για μια χώρα που σχετικά λίγε εξαγωγέ κάνει. Κατέβαλαν τι αμυγές προσπάθειε οι Βιετναμέζοι ε, για να εξελίξουν την ε, μεταποίησή τους και να την κάνουν και σύντονη μετά όσο εμείς ε, ζητούμε. Όσον αφορά το, τώρα τον Παγκάσιο, όντως, πήγαν εκεί οι συνάδελφοι, εξήτασαν τα πράγματα και δεν ήταν αρνητικά τόσο ανέφεραν, γιατί πρόκειται για ένα ψάρι το οποίο το, το, το, το καλλιεργούν όπως πρέπει και γίνονται και εξαγωγές όπως πρέπει. Υπάρχουν προβλήματα τιμολογιακής πολιτικής, είναι ανταγωνιστικό και αρέσει, δεν έχει κόκαλα. Οπότε και οι εστιατόρες επίσης το προτιμούν. Είναι πάρα πολύ κυστική η τιμή του, οπότε και αγοράζονται μεγάλες ποσότητες. Και οι πρωταθλητές στις αγωγές είναι η Ισπανία. Για μην έχουμε εργολικές αγωγές, υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας. Τα μέσα εμπορικής άμυνας. Και έχουμε έρθει σε επαφή με αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον ανταγωνισμό για το Παγκάσιο και μας ζήτησαν να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να κινητοποιηθούμε, να επικαλεστούμε αυτά τα μέτρα εμπορικής άμυνας, τα μέτρα αντιντάμπικα ας πούμε τις ρήτρες διαφύλαξης, ε, τα μετρα αντιντάμπινγκ. Ε, είμαστε ανοιχτοί. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα αυτά. Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε την εξέλιξη της αγοράς για το ψάρι αυτό. Και επίσης, στο Ανόη συνεργάζεται πάρα πολύ στενά η αντιπροσωπεία μας με τις πρεσβείες των χωρών μελών, της Ισπανίας, όπου βέβαια είναι και ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Αλίας και βρίσκεται και ως πρέσβης. Επομένως, παρακολουθούμε από κοντά τις εξαγωγές. Οι Βιετναμέζοι έχουν καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν κάποιες διαφοροποίησεις στις εξαγωγές τους και το ότι θα πρέπει να εξαγάγουν λιγότερο στην Ευρώπη και να κατευθυνούν περισσότερο προς Αίγυπτο, Περού, Βραζιλία Έχουμε μελέτε συγκεκριμένε πάνω σε αυτό και βεβαίω. Όποιο θέλει περισσότερε πληροφορίε θα του δώσουμε. Τώρα όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει για, τον, για την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική ακριβώς θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το οποίο είπε η Υπουργό το πρωί. Γιατί αποφασίστηκε η μεταρρύθμιση αυτή να ενταχθεί στην γενικότερη μεταρρύθμιση της ε, αλήθικης πολιτικής. Γιατί ακριβώς η κοινή οργάνωση αγοράς, σαν μεταρρύθμιση, θα πρέπει να περάσει με την γενικότερη μεταρρύθμιση της ε, αλήθικης πολιτικής. Βέβαια υπάρχουν εδώ πέρα θέματα στην ε, κοινή οργάνωση της αγοράς που αφορούν τις οργανώσεις των παραγωγών, όπου αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο παράγοντα, μεταβλητή για την μεταρρύθμιση. Δεν ωφελεί το να προχωρήσουμε προς μεταρρύθμιση χωρί και να έχουμε εν μέρη μεταρρύθμιση ενώ ταυτόχρονα ε, δεν έχουμε δει όλα τα μέτωπα τη γενικότερη μεταρρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε συζητήσει με τους εμπλεκόμενου και τα συζητούμε. Διότι έχουμε πει ότι το σύστημα υποστήριξής μας θα πρέπει να αναθεωρηθεί και αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να σταματήσουμε να ενισχύουμε από τις τσέπες των φορολογουμένων όμως είμαστε πρόθυμοι να δούμε πώς θα βρούμε κάποια πιο απλά μέτρα και μέσα γιατί σήμερα η νομοθεσία είναι πάρα πολύ πολύπλοκη ας πούμε για την αποθυματοποίηση των ψαριών εδώ να, να κάνουμε κάποιες ε, απλουστεύσεις. Είναι θέμα της, ε, του καλού χρονισμού της θέσης εμπορία των ψαριών. Έχουν πολλές ιδέες και προτάσεις που συζητούνται στα πλαίσια της γενικότερης ε, μεταρρύθμισης. Η Ισπανική Προεδρία θέλει να προχωρήσουμε, όμως δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Οπότε και αυτό το θέμα και τα άλλα θέματα της μεταρρύθμισης θα συζητούμε με τους εμπλεκόμενους. Τελεία εδώ, κυρία Πρόεδρε. Και υπάρχει άλλωστε ο παρακαθήμενος συνάδελφος. Κυρία Πρόεδρε, που ασχολείται με τα θέματα εμπορίου. Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μια επιπλέον ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι υπέρ του καθεστώτος ανταλλαγών μέσω των δασμολογικών ε, ε, τρόπων ή θέλετε να το αλλάξετε αυτό. Ε, vous parlez des quotas tarifaires, je Μιλάτε για ποσοστώσεις δασμολογικές. Όχι, όχι. Όχι, είναι μια μεταβλητή προσαρμογής. Γιατί χωρίς κανεί να πειράξει τους ε, δασμούς και τους τελεστές μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ε, εισαγωγές ε, κάνοντα κάποιε παρεκκλήσει στην φορολόγηση και έτσι κανονίζουμε να εισάγονται όσα ψάρια αντιστοιχούν στις ανάγκες της βιομηχανίας μεταποίησης. Άρα αυτό το μέτρο μάλλον μα εξυπηρετεί και πρέπει να, μην, ε, να μείνει, γιατί μπορεί να λειτουργεί ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και οι δασμοί. Ναι, ευχαριστώ. Μιλούσαμε με τον κύριο Στίβενσον και αφαιρέθηκαμε. Με συγχωρείτε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ο πρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Άμιλατ σας είπε λίγα πράγματα για μένα. Είμαι από τη Γενική Διευθύνση Εμπορίου. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και είμαι ευγνώμων που ο κύριος Κάντεκ ε, μας ενέπλεξε σε αυτή την ε, τόσο ενδιαφέρουσα, πολλά υποσχόμενη διαδικασία μέσω της ε, έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας του όπως και κάποιες άλλες γενικές ε, διευθύνσεις, το αποστήλαμε και εμείς στη δουλειά μας, ε, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη συνεισφορά μας, αλλά Έχω ήδη αρχίσει επαφή με τον κύριο Κάντε και, και με τον βοηθό του και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε σε προσωπική ε, επαφή. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου θα είναι εταίρος σε αυτή τη διαδικασία. Να πω ότι είναι μια μορφή πρωτοπορία αυτή η διαδραστηριότητα. Μετά από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχουμε νέε υποχρεώσει διαφάνεια, ε, οι οποίε μα επιβάλλονται βάσει του άρθρου 207 της συνθήκη. Υπάρχουν κάποιες ε, πολύ σημαντικές προκλήσεις ε, που προκύπτουν από αυτή τη διαφάνεια στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ε, οι πληροφορίες που διατίθενται και το πώς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως εμπιστευτικές ε, ή μη. Να σας ε, πω όμως ότι όπως είπε και ο κύριος Δεγκούχτ, ο υποψήφιος επίτροπος εμπορίου, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να ανταλλάσσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, ακόμα και εμπιστευτικά κείμενα θα μπορούσαν να δοθούν ε, αν τηρούνται κάποιοι κανόνες εμπιστευτικότητας. Ε, τα βασικά πράγματα, τις λεπτομέρειες εξετάζουμε ακόμα, εμπλέκονται αρκετές ε, γενικές διευθύνσεις επιτροπές, αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα τις χρειάζεστε τις πληροφορίες θα τις έχετε. Ως υπεύθυνο ε, τώρα της Γενικής Διεύθυνσης ε, Εμπορίου θα είμαι ε, υπεύθυνο για κάποιες πτυχές αυτού του φακέλου. Άκουσα και την έκθεση του ΠΟΕ που παρουσιάστηκε πριν από λίγο. Κάποιες από τις διαπιστώσεις της εκθέσεως ήταν ε, ευνοϊκές για μας. Για παράδειγμα, οι αλλαγές ε, που θα γίνουν σε θέματα απελευθέρωσης που προκύπτει από τις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι θα υπάρχουν όλο και λιγότεροι παραδοσιακοί δασμολογικοί φραγμοί και καλό είναι τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για την ε, περίοδο στην οποία θα μπορεί να προστατευτεί ο τομέας ε, με τη βοήθεια φυσικά και των κλασικών μέσων και από εκεί και πέρα να πω ότι τους στους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ να ετοιμάσουν τις συστάσεις για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Εμείς θα είμαστε εταίροι. Να επανέλθω τώρα σε αυτή την ε, ίδια πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολύ χρήσιμες συστάσεις ε, προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάντεκ για να ολοκληρώσουμε με το θέμα. Euh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ε, ε, συνεργασία και για την μελλοντική του συμβολή ε, δεν με πείσατε κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια των εισαγωγών από την Αποανατολή αλλά θα το ξανασυζητήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν, άκουσα τις παρατηρήσεις σας, είμαι στη διάθεσή σας για να ε, τις περιλάβω και εσείς θα με τροφοδοτήσετε με στοιχεία για την έκθεση. Η πρώτη ανταλλαγή δείχνει όμως ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ε, την ομίγυρη και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι το πολύ ενδιαφέρον ε, ε, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, οι βουλευτές σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάντε και ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρενέβη. Με αυτό ολοκληρώσαμε το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο 11 έκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίμακος προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης. Όπως γνωρίζετε, στην συνεδρίαση των συντονιστών το Σεπτέμβριο αποφασίστηκε να γίνει μια γνωμοδότηση επί του θέματος, οι σοσιαλιστές την ανέλαβαν και ο συντάκτης είναι ο κύριος Κρήτον Σένης Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σας δώνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα τα πω αγγλικά. Γιατί μπορεί να διευκολύνω με την ορολογία, λέει ο Γνωρίζουμε ότι οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών για την επόμενη 20 ετία ή 30 ετία έχουν ε, ήδη καθοριστεί βάσει των ε, εκπομπών μας. Ακόμα και αν σήμερα σταματήσουμε να εκπέμπουμε ε, αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου, οι αλλαγές θα είναι εμφανείς για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Βέβαια, αν δεν κάνουμε τίποτα, μέχρι το 2100 στο τέλος δηλαδή του αιώνα μας ε, είναι ελάχιστες οι να επιβιώσουμε σε αυτό το πλανήτη. Η θάλασσα είναι ο πιο σημαντικός αυτορυθμιζόμενος μηχανισμός ε, της αντιμετώπισης του κλίματος. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός μας σύμμαχος στην προσπάθειά μας και για να σταματήσει η αλλαγή του κλίματος και για να είναι ε, οι ποιότερες οι επιπτώσεις. Να σας δώσω μία εικόνα. Για παράδειγμα, αν αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα, ε, αυτό σημαίνει ότι στη Μεσόγειο θάλασσα και σε όλη την Νότια Ευρώπη η αύξηση θα είναι κατά 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Βόρειο Πόλο η αύξηση θα είναι κατά 16 βαθμούς Κελσίου. Ως προς το τους ωκεανούς, ε, σε γενικές γραμμές η αύξηση θα είναι γύρω στους 2 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ωκεανοί είναι αυτοί που θα επιτρέπουν η αύξηση να είναι μικρότερη από ό,τι θα ήταν σε άλλη περίπτωση. Η δυνατότητα απορρόφησης ε, άνθρακα και αλατός μας επιτρέπει να ε, αντιδράσουμε, μας δίνει περισσότερο χρόνο για να αντιδράσουμε στο φαινόμενο. Και ού μόνον αυτό, το 50% των αιτήσεων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου είναι απορροφούμενα από τα φυσικά οικοσυστήματα. Και υπ' αυτή την έννοια, οι περισσότερε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και των υπολείπων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου απορροφούνται από του ωκεανού. Αυτό βέβαια έχει κάποιε επιπτώσει για του ωκεανού. Υπάρχει κορεσμός ε, λόγω ε, άνθρακα. Το ωκεανικό pH αλλάζει και φυσικά όπως είπαμε και πριν η θερμοκρασία αυξάνεται. Μπορεί να βρεθούμε λοιπόν ενώπιον και ε, πιθανών αλλαγών στα θαλάσσια ρεύματα. Αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις και για τα αλλιευτικά αποθέματα και για τη θαλάσσια ζωή εν γέννη. Θερμότερες θάλασσες σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη απόσταση από την επιφάνεια. Είναι μικρότερο λοιπόν η επιφάνεια της θάλασσας στην οποία μπορούμε να έχουμε, η έκταση της θάλασσας στην οποία μπορούμε να έχουμε ε, ζωή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο ε, μικρότερη είναι η απόσταση από το βυθό της θάλασσας. Η θάλασσα λοιπόν κοραίνεται λόγω της ε, παρουσίας του άνθρακα και υπάρχει και κάτι επιπλέον. Μειώνεται η δυνατότητα απορρόφησης των ωκεανών. Επιστημονικώς ε, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι από το 2000 έως το 2007 η, πρόσληψη, ε, άνθρακα, η δυνατότητα συγγνώμη, πρόσληψης άνθρακα των ωκεανών μειώθηκε. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι θάλασσες φτάνουν στα όρια τους. Στο μέλλον λοιπόν Όσο περισσότερο οξύνονται οι ωκεανοί, πλήττεται η επιβέωση ε, αρκετών θαλάσσιων ζώων και των κορελογενών ζωνών. Οι κοραλιογενείς ζώνες στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου έχουν ε, είτε καταστραφεί είτε έχουν αποχρωματιστεί, έχουν ε, γενικώ υποστεί τεράστιες καταστροφές. Και ο ρόλος των κοραλιογενειών εφάλων στη ζωή των ε, θαλάσσιων όντων είναι υψής της Θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε ωκεανούς χωρίς ε, έμβια ζώα ή ε, κοραλιογενείς Φυσικά θα υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις και για την κοινωνία μας και για την οικονομία μας. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε βιώσιμα λιευτικά αποθέματα και τα αλλιευτικά αποθέματα εξαρτώνται όχι μόνο από, την, ε, από το επίπεδο αλλά και από τις επιτρό, ε, επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος, ε, ε, λοιπόν, και η αντοχή του κλίματος είναι πολύ σημαντική για να δούμε τι θα γίνει και με τα αλλιευτικά αποθέματα. Αν εφαρμόσουμε συγκεκριμένες αλλιευτικές τεχνικές, ε, σε περι... πολλές περιπτώσεις, ε, κυρίως της παράκτιας αλλίας, μπορούμε να διατηρήσουμε την ε, ισορροπία της θαλάσσιας διατροφικής αλυσίδας. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις, πιέσεις και στις παράκτιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρήπανση που θα προκύπτει από τις παράκτης δραστηριότητες και άλλες επιπτώσεις σε δραστηριότητες που γίνονται επεξηράς. Υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση, κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί καταλήλως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα την οικοσυστημική προσέγγιση, αυτή είναι η της σημασίας για οποιαδήποτε ε, πολιτική θέλουμε να ακολουθήσουμε και φυσικά αυτό συνάδει και με το στρατηγικό πλαίσιο για τις θάλασσες. Ένα ακόμα λοιπόν σημαντικό θέμα είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προκειμένου να ε, γίνουν οι ιδέωσες προσαρμογές και για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ολοκληρώνοντας να πω ότι θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε και τη δυνατότητα να έχουμε ένα κόσμο όπου οι παράκτης περιοχές θα είναι περιοχές τις οποίες τμήμα του εισοδήματος των αλλιέων θα ε, από δραστηριότητες ή ακόμα και επιδοτήσεις για δραστηριότητες οι οποίες θα αυξήσουν την αντοχή του κλίματός μας. Θα αυξήσουν τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τη γη μας από την αλλαγή του κλίματος και να μειώσουμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και για τα αλλευτικά αποθέματα και για τη ζωή εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρσένη. Ο κύριος Καντέκ έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση αυτή πολύ σωστά λέει ότι η κλιματολογική αλλαγή είναι αδιαφυσβήτηση και χρειάζονται μέτρα για να μειώσουμε τις επιπτώσεις και χαίρομαι διότι θα ενταχθεί ε, η βάση αυτής της προτάσεως η μάχη κατά των κλιματολογικών αλλαγών σε όλες τις πολιτικές ακόμη και τις αλληλίες γιατί επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και ε, χρειάζεται μία, ένα τέτοιο μέτρο. Ε, αυτό θα είναι το δεύτερο βέβαια, η δεύτερη φάση της εργασίας μας προς το παρόν όμως θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γίνουν ε, μελέτες για τις τάσεις που διαμορφώνονται κατόπιν της, της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας. Το ανέφερε ο κύριος κύριος αλλά τα αποτελέσματα θα πρέπει να μεταδοθούν επίσης και στην Επιτροπή και πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική αλληλεία στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι και θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της ε, θέρμανσης της ατμόσφαιρας και όχι μόνο η αλληλεία. Ε, δεν πρέπει να στιγματίζουμε την αλληλεία σε αυτό το τομέα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μιλάμε για υπεραλληλεία ε, στα αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή δεν πρέπει ουσιαστικά να θεωρήσουμε ότι ότι ε, η ε, αλληλεία ευθύνεται εκείνο από διοκομπομπέως τράγος ε, για την κατάρρευση των οικολογικών συστημάτων. Επίσης δεν νομίζω ότι αυθαίρετα πρέπει να μειώσουμε, το, να μειώσουμε τον αλληλευτικό στόλο αλλά να την ρυθμίσουμε καλύτερα. Μην ξεχνάμε τα άλλα πλοία και τις επιπτώσεις τους από πλευράς διοξιδίου του άνθρακος. Και στην παράγραφο 6 τέλος η εξοπλισμοί πρέπει να βελτιωθούν σε, όλα, σε όλους τους τόλους για να υπάρχει αηφόρος αλληλεία και η κυρία Δαμανάκη στο σημείο αυτό πρότεινε ενδιαφέροντες, ενδιαφέροντα μέτρα δηλαδή αλλαγή των μηχανών των υπαρχόντων πλοίων πρώτα σχόλια είναι αυτά και θα έχουμε ευκαιρία να ε, τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Δεν έχουν πολύ χρόνο. Παρά το ότι προσέχει την αυτή η έκθεση, αλλά όμω να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μακάρθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τόσο ακούσαμε σήμερα. Έχουμε σημειώσει πάρα πολλά στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά τη Λευκή Βίβλο, θα πρέπει να γίνει η Ευρώπη πιο αποτελεσματική στην αλλαγή του κλίματο εχουμε Έχουμε δύο ε, στάδια. Πρώτα-πρώτα η ευρωπαϊκή δράση και μετά εθνική. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τι παρακτές περιοχές για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Επίσης ε, έχουμε ένα συνδευτικό έγγραφο το οποίο ασχολείται με αυτά τα θέματα και εξηγεί τι μέτρα θα πρέπει να λεφθούν τόσο ώστε να είναι πιο εύκολη προσαρμογή. Σας ε, εγγυώμαι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προσαρμογή και τι αλλαγές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ούτω ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα. Ε, και αυτό όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο και όσον αφορά τη μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΠ. Το σχέδιο γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να λειτουργεί καλά η διαχείριση των παρακτήρων περιοχών και μεγάλη μου χαρά για να μπορέσουμε να έχουμε μακρόπνοη καλή ε, ε, στρατηγική αναφιωρούμε την σύσταση του 2002 και ήδη από πέρσι κάναμε μια μελέτη επιπτώσεων που θα γίνει και φέτος μαζί με δημόσια διαβούλευση τα οικοσυστήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και λέει σαφώς το, το, η Λευκή Βίβλος το, είναι οι επιπτώσεις τη αλλαγής του κλίματος. Οπότε, επ' αυτού έχουμε αυτό το πλαίσιο και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια στρατηγική προσαρμογής. Άρα θα είναι πάρα πολύ σωστό, ε, εάν συμφωνείτε, να θυγεί και η πτυχή υποφορά της θάλασσας. Βεβαίω και πρώτη θέμα θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ευχαριστούμε. Φράγκα. Σας ευχαριστώ. Θέλετε το λόγο σχετικά με αυτό. Όχι. Ε, τότε να τελειώσουμε αυτό και αν δεν σας πειράζει μετά να μιλήσετε. Κύριε Αρσένη, θέλετε το λόγο. Προθεσμία για τροπολογίες. Είναι η Τετάρτη, Δευτέρου, το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στις 23. Κυρία Λέβιν. Αν γίνεται, είναι διαδικαστικό, να κοιτάξουμε την επαφή μας για να μας συμβουλεύσουν νομικές υπηρεσίες για το τι γίνεται με το Μαρόκο. Αυτό το σημείο της διάταξη και αν είναι δυνατόν. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτήν την ε, νομική γνωμοδότηση πριν τελειώσει η συνάντησή μας γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την συνεδρίαση που θα φορά ακριβώς το θέμα αυτό. Ναι, αλλά δεν μας μένει χρόνος, έχουμε την έκθεση Φερέιρα που είναι εδώ. Είναι κατεπήγον. Και χρειάζομαι και λίγη ώρα για να τα ψηφίσουμε. Αλλιώς να το αναβάλουμε το θέμα για την επόμενη συνάντηση. 12 το σημείο χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. Τροποποίηση κανονισμού 708 κάθετο 2007. Η εισηγητής είναι ο κύριο Φερέιρα. Εδώ έχει αλλάξει η νομική βάση όταν άρχισε να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ο κύριο Φερέιρα είναι ο εισηγητής. Αλλά δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέσσερα λεπτά maximum.